Good evening. Good evening. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Evening, ladies and gentlemen. Do you have your... Λοιπόν, έχετε τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε. Σας παρακαλώ. Όχι, τι όχι. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε τις κάρτες στα μηχανήματα. Είστε έτοιμοι. Completely. Let us start then. First, Πάμε λοιπόν. Πρώτα θα ψηφίσουμε δοκιμαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι, χαίρεστε που ψηφίζετε Δευτεριάτικα 7 ώρα το βράδυ στο Στρασβούργο. Γι' αυτό ψηφίζουμε τώρα, παρακαλώ. Πέρασε. Α, Μισό-μισό. Ε, δεν τρελαίνεστε κιόλα, αλλά δεν είναι σαφέ. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, να ζητεί κανεί. Όχι, καλά. Ε, αγαπητοί φίλοι, έχουμε πολλή δουλειά σήμερα και πολλέ ψηφοφορίε. Έχουμε και τις... Κοιτάξτε κατάλογοι ψηφοφορίας. Είναι τόμος εδώ πέρα. Να οργανωθούμε και να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ε, πρώτη έκθεση που έχουμε να ψηφίσουμε. Εισηγήτρια είναι η κυρία Πιλάρ Ντελ Καστίγιο, Ευρωπαϊκός Κώδικας Ελεκτρονικών Επικοινωνιών, αναδιατύπωσης. Πάμε. Αρχίζουμε αμέσως να ψηφίζουμε, παρακαλώ. <clears throat> Τροπολογία 145. Ψήφι υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασε. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία και τελειώνει. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογικός είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 296 και 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 297 και λίμπε 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 441 λίμπε και 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίζουμε τη 298 ηλεκτρονικά πέρας. Εγκρίνεται. 317 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 318 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 3, Α, έλεγχο θέλετε για τη 16 της Λίμπε. Παρακαλώ. Λίμπε 16, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Στο ΕΛΚ είστε ένας υπεράριθμος. Απορρίπτεται. 3.19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 320 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 322 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ. 322. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 324 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 325 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 327 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 79 το πρώτο τμήμα ορίστε α μόνο το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Compromise 7 in favor. Η 7 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στη σελίδα τώρα υπαριθμών 9. Από 94 επισημένο. 9. Η τροπολογία 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ τσεκ φωνές. Καλά. Να σηκώνετε και χέρια όμως τι τσεκ. Λοιπόν, 37. Το τσεκάρουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Στο ΕΛΚ ένας υπεράριθμος. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια συνάδελφοι. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 38. 38 πέρας. Εγκρίνεται. 396 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Μερικές τροπολογίες στη συνέχεια, όπως βλέπετε, τις βλέπετε μαζί, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Επόμενη ενότητα υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να διαβάζω όλες τις τροπολογίες, τώρα τις βλέπετε. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά απόχες εγκρίνεται. Ωραία, θέλετε έλεγχο, παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 39 πέρας. Εγκρίνεται. 406 και 407 επέ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 408 επέ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 409 και 410 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 411. Λίμπε 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 412 και 21 της Λίμπε μαζί. Καθώς και η 413 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4.14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4.15 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Ελέγχουμε την 4.15. Τι θα γίνει με το ΕΛΚ. Έχετε έναν παραπάνω. Όχι πέρας. Όχι ακόμα. Έχετε λίγη ώρα ακόμα. Να βγάλετε από το ΕΛΚ μία κάρτα παρακαλώ. Μήπως εγώ. Καλώς. Εγκρίνεται. 416 και λίμπε 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επαληθεύουμε λοιπόν τη συμβαστική παριθμό 3 ηλεκτρονικά. Το ΕΛΚ εξακολουθεί να έχει ένα παραπάνω που ψηφίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Τι σελίδα είναι, ρωτάει κάποιος. 15. Ε, συμβαστική 2 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται η συμβαστική 8 στη σελίδα 17. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 21. 496 και κουλτ 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 5. Και 497 τι έγινε. Α, sorry. 497 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Α, δεν κοιμάστε καθόλου, σας δοκίμαζα. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές αυτή θέλει έλεγχο γιατί είναι και συμβαστική. Ε, συμβαστική 5. Α, τώρα είναι σαφές, προηγουμένως δεν ήταν όμως. Πέρας. Σας παρακαλώ να σηκώνετε χέρια. Πάμε σε λίδα 24, συμβαστική 9α. Ηλεκτρονικά, κατευθείαν, γιατί σίγουρα θα είναι πολύ σφιχτή. 9α. Πέρας. Εγκρίνεται. Καλώς αφού εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 10. είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. είπε. Συγγνώμη. Σελής 28. Α, έχουν διαφορετική ρύθμιση οι κατάλογοι ψηφοφορίας. Λοιπόν, σταματάω να λέω σελίδες. Ζητάω συγγνώμη, αλλά τι να κάνω. Συμβαστική 11. In favor. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 563 και λίβε 25 και ΙΜΚΟ 96 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 564 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 564. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πάτε 6-7 σελίδες πιο κάτω. Σας παρακαλώ. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15-20 σελίδες πιο κάτω τώρα. Στο δικό μου κείμενο είναι σελίδα 47, συμβαστική 1. Περιμένω να το βρείτε. Ε, Συμβαστική ένα. Δεν σας αφήνω καθόλου σε χλωρό κλαρί να κοιμηθείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμβαστική παριθμόν 1. Compromise, compromise Συμβαστική παριθμόν 1. Δεν ξέρω τι σελίδα έχετε. Ωραία. Η συγγήτρια. Έχει πάντα δίκιο. Λοιπόν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άλλες 18 σελίδες κάπου εκεί πιο κάτω. Πάμε στη συμβιβαστική 12α. 12α. Yes, I Δεν αρχίζει κανείς, δεν ψηφίζει κανείς. Περιμένω. Χρόνο έχουμε, άπλετο. Λοιπόν, συμβιβαστική 12α, είναι στη σελίδα 70. Είστε έτοιμοι. Ωραία. Ηλεκτρονικά θα την ψηφίσουμε αυτή. Γιατί θα είναι πολύ μικρή η διαφορά. 12α. Πέρασα. Εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. 13α. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τη συμβαστική 13α. Εγκρίνεται. Τι έγινε, τρέχει τίποτα. Θέλει κανείς να πει τίποτα. Όχι. Καλώς. Προχωρούμε λοιπόν. Αρικές σελίδες πιο κάτω. 7-8 ξέρω εγώ. Η ε, συμβιβαστική Τώρα να σας πω ποια είναι η συμβιβαστική, δεν ψηφίζω ακόμα. 1066D. d Δεν είναι συμβαστική, είναι η τροπολογία κανονική στη σελίδα 76. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 1066D. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ήμκο 157 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Δυστυχώς χρειάζεται και πάλι. Για την 157. Άρχεται και κλείνει. Εγκρίνεται. 1067 ψήφι υπέρ. Κατά. Και εδώ χρειάζεται επαλήθευση. 16. 1067. Πέρας. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Στην τροπολογία 1072. 1072. Διαφωνεί κανείς με την προφορική τροπολογία αυτή. Όχι. Ωραία. Προτείνω το εξή τώρα. Για το πώς θα ψηφίσουμε. Σας παρακαλώ να με ακούσετε. Ε, είμαστε στην τροπολογία 1072 που θα την ψηφίσουμε μαζί με την προφορική που συνεχίζεται και στην επόμενη σελίδα μαζί με την 160 της ΙΜΚΟ. Και μετά θα ψηφίσουμε την τροπολογία 1071 σε περίπτωση που δεν εγκριθεί. Εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει, υπάρχει συμφωνία να ψηφιστεί έτσι. Η 1072 μαζί με την προφορική και μαζί με την 160 της ΣΥΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει η άλλη. Μάλλον όχι. Ναι, και ψηφίζουμε τη 1073. Υπέρ. Κατά. Και τι έγινε η 1071. Κατέπεσε. κατέπεσε εφόσον εγκρίθηκαν οι δύο άλλες. Εφόσον υπερψηφίσαμε την 160 της ΣΥΜΚΟ και τη 1072, η 1071 καταπίπτει. Καλώς. 1073 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. Δύο τροπολογίε 1074 και ΜΚΟ 161, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1075 και ΕΜΚΟ 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1076 και ΛΥΜΠΕ 43 και ΕΜΚΟ 163. Όχι. Όχι, όχι. Οι δύο προηγούμενε μόνο. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. ψηφία Ισοψηφία. Απορρίπτεται. Ήμκο 163 Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα θα πάμε λίγο πιο κάτω. 6-7 σελίδες πάλι. Θα περιμένω να γυρίσετε τις σελίδες σας. 148 λίμπε. Δεν θα ψηφίσουμε ακόμα. Είναι σελίδα 85. Μαζί. Με άλλες τροπολογίες. Λοιπόν, 148 λίμπε 1, 149 λίμπε 2, 150 λίμπε 3. Όλα αυτά μαζί. Ομού, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 151 και ΙΜΚΟ 1 μαζί είπε κατά έλεγχος παρακαλώ καλύτερα εγκρίνεται 152 και λίμπε 4 υπέρ κατά και αυτό θέλει έλεγχο 152 και λίμπε 4 πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα, τέσσερις τροπολογίες μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Η 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήμικο 4, τμήμα πρώτον, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμικο 5 υπέρ, κατά απορρίπτεται. Καλά και αποχές ξέχασα να πω, αλλά απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά αυτό χρειάζεται απολύθευση. 169 παρακαλώ. Απορρίπτεται. 170 και λίγο 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΛΥΜΠΕ 6 υπέρ κατά εγκρίνεται έλεγχο θέλετε παρακαλώ ΛΥΜΠΕ 6 επαληθεύουμε αυτή την τροπολογία πέρας εγκρίνεται 176 υπέρ κατά έλεγχος 176 πέρασε απορρίπτεται 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για πάμε παρακάτω τώρα στην τελευταία σελίδα Αν μπορείτε ακόμα να βρείτε την τελευταία σελίδα. Διότι είναι η τελική ψηφοφορία για την ε, σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Με ονομαστική κλίση. Είστε έτοιμοι πιστεύω. Πάμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται η έκθεση με συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία Καστίγια. Έχουμε και άλλη ονομαστική ψηφοφορία για να αρχίσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 69 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και πάλι με τεράστια πλειοψηφία για να αρχίσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και συνεχίζουμε. Α, κυρία εισηγήτρια, βεβαίως. Ε, χωρίς ε, μικρόφωνο. Και αγαπητέ Πρόεδρε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλα τα θέματα είναι σημαντικά, αλλά για το θέμα αυτό θα ε, έχουμε καθοριστική επιρροή ε, για το μέλλον στην Ευρώπη, των υποδομών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τώρα θα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα για να δώσουμε συνέχεια και να είμαστε συνεπείς στα όσα ψηφίσαμε σήμερα, έτσι ώστε να έρθει σε αίσιο πέραση η απόφαση και ο κανονισμός στην Ευρώπη για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για να βελτιώσουμε τη διασύνδεση και τη συνδεσιμότητα, όπως λέγεται τώρα, που είναι το σημαντικότερο. Βεβαίω είναι και τα δικαιώματα των καταναλωτών και η εσωτερική αγορά. Σήμερα όμως αυτό που θα ήθελα να πω είναι να σας ευχαριστήσω όλους και τους κοιόδες συγητές και τους υπαλλήλους. Δυστυχώς η ομιλήτρια δεν ακούγεται, δεν μιλάει στο μικρόφωνο. 1.154 ήταν οι τροπολογίες και πάνω από 1.000 καλύφθηκαν από τους συμβασμούς. Ξέρετε ότι έχω και ειδικό βοηθό για αυτό το θέμα και θέλω να τον ευχαριστήσω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και τη βοήθεια τη γραμματεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. uh, we ε, δεν θα ξεκινήσει τώρα μια συζήτηση, αλλά θέλετε να πείτε ναι. Εκ μέρου των σκιωδών ευχαριστώ τη συγκίτρια. Ήταν πολύ σκληρή δουλειά, πολλέ τροπολογίε, πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να συγκρίνω. Όταν δουλεύει και δεν έχει σύνδεση, είναι το ίδιο. Αν δεν πετύχουμε αυτό, η Ευρωπαϊκή Σύνδεση θα διασπαστεί. Ξέρουμε πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό το θέμα. Μπορεί να καθίσουμε μέχρι τι 12 να το συζητάμε, αν το ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, φίλοι, ας πάμε στην πρόταση για ε, τον Φορέα Ευρωπαίων, Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τι ηλεκτρονικές επικοινωνίε. Ε, Ευγέννη Τόσονόφσκι, ο, ο εισηγητη 1, 2, 19, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε την σελίδα πριν από την τελευταία σελίδα. Όλο μαζί λοιπόν, περίπου 60, 60 σελίδες, ο κύριος Τοσιονόφσκι μας έχει ε, δώσει κάτι το ξεχωριστό για απόψε. Η πρώτη τελευταία σελίδα λοιπόν, ή ακόμη και η τελευταία, δεν ξέρω. Τοπολογία 163 υπέρ, κατά, ξανά, γιατί κανείς φαίνεται να μην θέλει να ψηφίσει. 1,63. 163 υπέρ, κατά. Επαλήθευση. And I close the vote. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές όχι να περίπλοκο. Ψηφίστε με ξεκάθαρο τρόπο. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 164. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Έχουμε έναν ΕΛΚ υπεράριθμο. Και πάλι... Ναι, την έχω αφαιρέσει εγώ. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Να το ελέγξουμε. 168. Επαλήθευση της ψηφοφορίας. Και πάλι ένας ΕΛΚ υπεράριθμος. Από το ΕΛΚ έχουμε έναν υπεράριθμο. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Για το σχέδιο της έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. I close the vote. Πέρα στις Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή και ε, δεύτερο ε, ψηφοφορία ε, σύμφωνα με τον κανόνα 69 ονομαστική ψηφοφορία για διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις. Άρχεται ψηφοφορία πέραση ψηφοφορίας. με συντριπτική ε, πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Ε, Ο εισηγητής θέλει να πάρει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους συναδέλφους, τους βοηθούς, η συνεργασία ήταν άψογη και κατορθώσαμε να οργανώσουμε όλες τις τροπολογίες σε μία. Ωραία, πάμε τώρα στην, στο τρίτο κατάλογο ψηφοφορίας. Ε, η συνάδελφος Κάλλας είναι η σύγκριτη. Ο σεβασμός ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και κατάργηση της οδηγίας ε, του παρελθόντος Τροπολογία 118 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 τροπολογίες συνολικά από το 120 μέχρι το 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 121 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνονται. 122 και 123 υπέρ. Κατά. Αποχές απορριπτονται. 128 υπέρ. Κατά. Ας την επαληθεύσουμε. 128. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 131-132 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε και αυτές. 131 και 132. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορριπτώνται αυτή τη φορά. 133 και 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Ας την επαληθεύσουμε. 137. Παληθεύουμε την 137 πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 138 και 64 υπέρ. Κατά. Ας την επαληθεύσουμε. 138 και 64 επαληθεύσει. Πέρασε της πληροφορία. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά ας την επαληθεύσουμε 143 άρχεται η ψηφοφορία Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται 145 μάλλον 144 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 τώρα υπέρ κατά Αποχές πρέπει να την επαληθεύσουμε την 145. Πέραση της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. 146 και 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά αποχές απορριπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μερικές σελίδες πιο πέρα. Συμβιβαστική 15. Κάποιες σελίδες προχωρήστε πιο κάτω. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 4-5 σελίδες προχωρήστε. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2-3 ε, σελίδες πιο κάτω. 2-90 υπέρ Κατά. Ας την επαληθεύσουμε. Πιθανό να, έχει, ε, να απορριφθεί. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 291 υπέρ. Κατά. Ας την επαληθεύσουμε. 291. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 302 εγκρίνεται. 303 υπέρ κατά αποχές. Α την επαληθεύσουμε. 303 επαληθεύση. Πέρσι ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 304 υπέρ. Κατά. Αποχέ. α την επαληθεύσουμε. 304. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 333, δεύτερο τμήμα. ψηφίσμα υπέρ. Κατά. Ας την επαληθεύσουμε. 333, δεύτερο τμήμα. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 343 υπέρ. Κατά. Ας την επαληθεύσουμε. 343. Επαλήθευση πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 344 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 346 υπέρ. Κατά. Ας την επαληθεύσουμε. 346 επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 348 υπέρ. Κατά. Εποχές ε, απορρίπτεται. 349 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ναι, απορρίπτεται. 350, 51 μαζί, υπέρ, Κατά. Α, την επαληθεύσουμε, ας την επαληθεύσουμε. 350 και 351 μαζί. πέραση η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 352 είπε Κατά. Ας την επαληθεύσουμε και αυτήν. 352. Πέρασε η ψηφοφορία.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 Αποχές και απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Ας την επαληθεύσουμε. 54. Επαλήθευση της 54. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Ας την παληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 65. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Ας την επαληθεύσουμε. Την 67. Επαληθεύση της 67. Και πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές, ας την επαληθεύσουμε. 69. Επαλήθευση για την 69. Εντάξει, εντάξει. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 75 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά Ας την επαληθεύσουμε. Την 82. 82 επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορριπτέται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά την 109 θα επαληθεύσουμε επαλήθευση της 109 πέρας της πληροφορίας απορρίπτεται Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 115. Ε, επαλήθευση τότε της 115. Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, απορρίπτεται. 116 υπέρ κατά. Θα την επαληθεύσουμε και την 116. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Συντριπτική πλειοψηφία, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Καλώς, not fair. Okay. Okay. Ωραία. Και τώρα περνάμε στην, στον ε, κύριο Πώς πρόταση όχι. Για τη συγκρότηση κοινή επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων. Έχουμε εννέα τροπολογίες συνολικά στην αρχή. Θέλετε, έχετε μάλλον αντιρρήσει να τις ψηφίσουμε όλες μαζί αυτές τις εννέα τροπολογίες που είναι στην αρχή του κειμένου υπέρ, κατά, αποχές, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Απορρίπτονται. Τροπολογία παριθμών 1. Ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 10. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Κόντα 1. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή κοκομπού 2 κοντ 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή κοκομπού 3 υπέρ συμβιβασμός 2 καταρχάς συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή κοντ 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή κοντ 4 υπέρ κατά. Το ελέγχουμε ηλεκτρονικά το σημείο αυτό. Κοντ 4. Έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚΑ. Δεν ψηφίζω εγώ. Κάποιος άλλος. Εγώ δεν μπορώ ούτως ή άλλως. Ποιος άλλος όμως ψηφίζει που δεν πρέπει. Α, μάλιστα, τέλεια. Μια χαρά είναι, μου λένε. <laughs> Πολλαπλασιαζόμαστε εδώ, ε. Κλανοποιούμαστε. Καθήμενοι. Α, απορρίπτεται. Rejected. Απορρίφθηκε η κοντ 4. 14. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κοντ 5 υπέρ, κατά, την ελέγχουμε ηλεκτρονικά την κοντ 5. Πέρας ΦΟΦΟΡΙΑΣ απορρίπτεται. Τώρα, συμβιβασμός 3, υπέρ. Κατά άποχες δεκτή. Τέσσερις τροπολογίες μαζί. Αντιρρήσεις δεν υπάρχουν. Υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Γίνεται αποδεκτή. Και τώρα περνάμε Α, ξέχασα να πω συγχαρητήρια. στον κύριο Και τώρα πάμε στο Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018. Το προηγούμενο ήταν το Omnibus. Τώρα μιλάμε για το οικονομικό έτος 2018. Γενικός προϋπολογισμός. Πρώτη τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποδεκτή. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά ελέγχουμε την 6 ηλεκτρονικά πέρας υποφορίας απορρίπτεται 7 υπέρ το πρώτο τμήμα υπέρ κατά άποχες. Ελέγχουμε και αυτήν ηλεκτρονικά, την 7. Το πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα της 7. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. Γιατί δεν υιοθετήθηκε το πρώτο τμήμα. 8. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 11 ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός αν υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτός. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμό 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτός. 23 υπέρ. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές δέκτη τελική ψηφοφορία με δομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας, δεκτή, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρα, πολυ παρακαλω να παραμείνουμε στην αίθουσα, γιατί έχουμε τώρα την τακτική, έχουμε τη συνεδρίαση μάλλον της Επιτροπής μας, παρακαλώ μείνετε στην αίθουσα.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 Uh, αγαπητοί... συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αγαπητέ κύριε Νίκα και υπόλοιποι, σας παρακαλώ, εάν θέλετε να συζητήσετε το οτιδήποτε, σας παρακαλώ έξω από την αίθουσα. Λυπάμαι που το λέγω, αλλά τώρα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ο κύριος Πουτικόφερ είναι ο εισηγητής. Όχι κυρία Μινκόφσκαγια, Μπιενκόφσκαγια, που θα έρθει επόμενα μέσα στα επόμενα 30 λεπτά. Τώρα είναι ο κύριος Μπουτικόφερ. Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο. Το σημείο 9 της διάταξης. Είναι μια γνωμοδότηση της ΣΥΤΡΕ για την έκθεση πρωτοβουλίας της ΙΝΤΑ. Okay. Um, on behalf, I understand, on behalf of Mr. Εκ μέρους του κύριου Μπουτικόφερ. Ο κύριος Τούρμες από τους Πράσινους. Θα την παρουσιάσει. Ο κύριος Μπουτικόφερ είναι στην Ορλομέλεια. Δυστυχώ δεν μπορεί να είναι και εδώ. Πρέπει να τη συζητήσουμε όμω τώρα, γιατί αλλιώ η ψήφο μα θα φτάσει πολύ αργά στην ψηφοφορία της ΙΝΚΟ. Όλοι οι σκιώδες, έχουν τα σημεία του κύριο Μπουτικόφερ, ε, τα εννέα σημεία, δεν θα τα διαβάσω, δεν βοηθάει. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση και ίσως συνεχεία Μπορεί να έρθει και ο κύριο Μπουτικόφερ ε, για να μας πει για κάποια τελικά συμπεράσματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο σχέδιο συγκεκριτή του ΕΛΚ, Ο κύριος Άντο Πατριτσέλο έχει το λόγο. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μπουτικόφερ, για το θαυμάσιο κείμενο που συνέταξε. Η ολοποίηση μιας ενιαίας αγοράς ψηφιακής φύσεως είναι ουσιαστική, ούτω ώστε να επιτρέψουμε στην Ευρώπη να παραμείνει μεταξύ των πρωτοπόρων της, της παγκόσμιας οικονομίας, στηρίζοντας και την αύξηση των ευρωπαϊκών εταιριών σε διεθνές επίπεδο. Το ίντερνετ και νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει ριζικά τις συνήθειές μας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες και η οικονομία. Είναι επομένως απαραίτητο να έχουμε μία όλο και πιο ψηφιοποιημένη αγορά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα εργαλεία, ούτω ώστε να εγγυηθούμε μία ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς εμπόδια και να εξασφαλίσουμε με ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και των καταναλωτών αλλά και των ατόμων γενικά. Πολλά από, τα εμπορικά, από τους εμπορικούς κανόνες δεν αντικατοπτρίζουν αυτή την πραγματικότητα που ζούμε. Οι κυβερνήσεις παντού βλέπουν ότι η παγκόσμια αγορά είναι όλο και πιο αλληλένδετη, οι αγορές μάλλον, και δημιουργούνται έτσι πλεονεκτήματα και για τις ε, ε, εθνικές εταιρείε, οι οποίες μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει τον ψηφιακό προστατευτισμό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ε, τον νομοθετικό κατακαιρματισμό και την, ε, τις γραφειοκρατικές τροχοπέδες να δημιουργήσουν προσκόμματα σε μια αγορά που εκτιμάται να βρίσκεται στα 415 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερε υπηρεσίε, με καλύτερε τιμέ, θα έχουμε περισσότερε επιλογέ και θα έχουμε νέε δυνατότητε απασχόληση. Η ψηφιακή αγορά μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίε για τι νέες, τι νεο, τις ε, και να επιτρέψει στις υπάρχουσες ε, επιχειρήσεις να απτυχθούν περαιτέρω μέσα σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τώρα, για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις πληρωμές online, η, η κατάρρευση των εμποδίων μπορεί να είναι μια ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης φιλόδοξη, ούτως ώστε να, να δημιουργήσει απτά ε, ωφέλη στους καταναλωτές. Είναι ουσιαστικό όμως να υλοποιήσουμε μια κοινοτική στρατηγική η οποία θα μας θα εγγυά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μια ισότιμη πρόσβαση στις ε, αγορές των τρίτων χωρών, ούτως ώστε να υπάρχουν απτά ωφέλη για τους καταναλωτές και να είναι σε θέση να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων και να ε, προωθήσει τους παγκόσμιους κανόνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά τον εισηγητή για το κείμενό του. Είμαι σίγουρος ότι χάρη στην σημερινή συζήτηση και χάρη στις προτάσεις που θα, θα κάνουμε μαζί τους ε, συναδέλφους και τις προτάσεις που θα κάνουμε μέσω των τροπολογιών που θα παρουσιάσουμε μέχρι αύριο θα φτάσουμε στο τέλος των διαπραγματεύσεων σε μια κοινή θέση και αρκετά φιλόδοξη ούτω ώστε να δώσουμε χρήσιμα στοιχεία στην Επιτροπή Δημοσι... Ε, Διεθνούς Εμπορίου, την Επιτροπή ΙΜΚΟ δηλαδή. Ευχαριστώ. Thank you very much, colleague, for your remarks. Ευχαριστώ Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις από τους σοσιαλιστές. Ο οποίος Κολουμπάτσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπιουτικόφερ για το έργο του στο θέμα αυτό. Χαίρομαι που ο προλαλής σας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον προστατευτισμό. Είναι διαφορετικές οι πρακτικές Υπάρχει ο γεωγραφικός αποκλεισμός, ε, υπάρχουν διάφορες πολιτικές, διάφορες τεχνολογίες, ε, περιπλοκή στην ε, προσφορά εναλλακτικών πλήρωμων. 22 μέτρα έχει εντοπίσει μια βελγική τράπεζα που επιβάλλουν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη για τη μεταφορά δεδομένων στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε τι θα γίνει αν αυτό συμβεί εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε ποια είναι τα εμπόδια για το ψηφιακό εμπόριο και να το καταργήσουμε. Τα, τα εμπόδια. Το ε, ψηφιακό εμπόριο και η ψηφιακή αγορά καλπάζει, αλλά διασυνοριακά είναι πολύ μικρό το κλάσμα σε σχέση με το σύνολο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αναπτυχθούν. Ε, πέρα από την τοπική αγορά, υπάρχει περιφερική, εθνική και διεθνής μέχρι και παγκόσμια με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Προφανώς χρειάζεται διεθνή συνεργασία ε, στην προστασία των καταναλωτών, στην μεταφορά και παράδοση δεμάτων και ε, στο ηλεκτρονικό εμπόριο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των τελωνίων για να μπορούμε να έχουμε καταχώρηση των ε, δικαιολογητικών και των φορτωτικών και των διαφόρων διασαφήσεων ηλεκτρονικά έτσι ώστε να καταβάλουν ηλεκτρονικά και τα τέλη και δασμοί. Έτσι θα μειωθεί το κόστος και θα είναι προς όφελος των διεθνών καταναλωτών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εργαστεί και σε ένα σήμα εμπιστοσύνη ψηφιακό και ηλεκτρονικό που να εξασφαλίζει ίδιους κανόνες και ίσους κανόνες παιχνιδιού για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πλατφόρμες αλλά όχι γενική υποχρέωση για τον ελεγκτή και για το μεσάζοντα ε, εκ των προτέρων. Θα πρέπει όμως να είναι εγγυημένα τα πνευματικά δικαιώματα και να ελέγχεται την περιεχόμενο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Βεβαίως δεν είναι ο μόνος τρόπος συνεργασίας αυτός για την ψηφιακή αγορά. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπογράφει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τρίτες χώρες, θα πρέπει να έχουμε και ένα κεφάλαιο για την ψηφιακή αγορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο ε, τύπου Σιγκαπούρης, Καναδά και τέτοιες συμφωνίες. Ενώ, ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μπαρέκοφ από το ECR, παρακαλώ. Η ψηφιοποίηση του διαδικτύου και οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν πολύ τις κοινωνίες μας, την οικονομία μας. Οι παραδοσιακές βιομηχανίες ψηφιοποιούν όλο ένα και πιο πολύ την παραγωγή και τις υπηρεσίες. Οι μικρότερες εταιρείες μπορούν να φτάσουν στους πελάτες τους ε, με ταχύτερους ρυθμούς και χαμηλότερο κόστος. Σήμερα ε, πολλές από τις οδούς εμπορίου δεν ακαλύπτουν αυτή την πραγματικότητα. Στο μεταξύ οι κυβερνήσεις δημιουργούν φραγμούς ε, που φράσουν την πρόσβαση στις αγορές ε, ή δημιουργούν ε, αθέμητα προλεκτήματα που δεν διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν αγορές online και θα πρέπει να καταργηθούν οι φραγμοί στο εμπόριο. Αυτό θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής διασφάλισης ε, μιας πρόσβαση πρόσβασης, θεμητής πρόσβασης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες είναι κλειδί. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ 1,7 τρισεκατομμύρια εκατομμύρια ε, ευρώ αξίας ε, προϊόντων στον κόσμο. Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στοχεύει στο να καταργήσει τους φραγμούς εμπορικούς χωρίς να μειώνει τις αξίες και την προστασία μας. Έτσι, η κυριότερη έμφαση είναι στα εξής. Τα μέτρα, στα μέτρα που περιπλέκουν το γενικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, τις απαιτήσει για τοπικό περιεχόμενο, τις φραγμούς στις επενδύσεις, ε, στην επιβράδυνση των διαδικασιών που ε, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ε, εταιρείε. Η ποιότητα του ψηφιακού δικτύου, η ταχύτητα του διαδικτύου και η διασυνδεσιμότητα θα επηρεάσουν τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων, τη διαφοροποίηση του προϊόντος που θα έχει θετικό αποτελεσμό για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Ε, από τους φιλελευθέρους η κυρία Βίλρικ. Ο κύριος Ντομινίκ Ρικέ είναι κανονικά ο σκιώδης Το μικρόφωνο αυτό δυστυχώς δεν λειτουργεί. Καλά πρέπει να πάρει κάποιο άλλο εμιλήτρια. Δεν θα μιλήσει η ομάδα των φιλελευθέρων. Okay. Καλώς. Επόμενη. Η κυρία Τόια, αντιπρόεδρός μας. Ευχαριστώ. Μόνο να προσθέσω κάνα δύο παρατηρήσεις. Νομίζω ότι η πρόταση του κυρίου, πρόταση του κυρίου Μπουτικόφερ είναι πολύ προσεκτική, πολύ ευρεία, όπως πάντα. Εγώ προσωπικά θα τόνιζα μόνο δύο σημεία. Πρώτον, ενώ εμείς προσπαθούμε να αναπτύξουμε το διεθνές εμπόριο, το ηλεκτρονικό πώς, το οποίο λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο που ξεπερνά τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει παράλληλα να έχουμε και κοινοτικά εργαλεία κατάλληλα. Εγώ θα μιλούσα και για την ανανέωση οδηγίας e-commerce, ηλεκτρονικό εμπόριο. Ε, γιατί εκείνος μιλάει για το παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για μια ενίσχυση, όπως είπε. Το είπε και κάποιο σε μια παρέμβασή του, ο κ. Πατριτσέλο για μια ενίσχυση του κοινοτικού πλαισίου. Συμφωνώ με αυτό. Δεύτερον, επίση υπάρχουν τρία πράγματα που μα απασχολούν. Οι επιχειρήσει, οι επιχειρήσει ε, που δίνουν ε, υπηρεσίε, ε, πέρα από τι επιχειρήσει που παράγουν αχαθά, οι καταναλωτέ και οι εργαζόμενοι. Εμά ω Επιτροπή μα ενδιαφέρει κυρίω το θέμα των επιχειρήσεων, το οποίο όμω δεν είναι ανεξάρτητο από την εργασία. Έτσι. Εγώ τα θεωρώ αυτά τα δύο αλληλένδετα. Θα ήθελα να σα πω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να αναπτυχθεί ένα εμπόριο, ψηφιακό εμπόριο, το οποίο σέβεται και τον εργαζόμενο. Όπως ξέρετε, διάβασα εδώ πέρα ένα άρθρο σε μια Ιταλική εφημερίδα, ότι υπάρχει το εξή φαινόμενο. Ε, υπάρχει ένας τρόπος εργασίας στους πιο παραδοσιακούς τομείς, ας πούμε, της ε, γεωργίας, όπου ε, υπάρχει απόλυτη εκμετάλλευση του εργαζόμενου. Δυστυχώς, με βάση έρευνες, ε, βλέπουμε ότι εκμεταλλευόμαστε απόλυτα και τον εργαζόμενο που εργάζεται στον ψηφιακό τομέα. Θα ήταν κρίμα να προχωράει έτσι η τεχνολογία, να προχωράνε οι δομές, να προχωράει η, προχωράει η άμυνα του καταναλωτή και όμως εμείς να αφήνουμε ε, τους παραδοσιακούς τομείς ας πούμε στο έλεος τους ε, και αύριο μεθαύριο και τον ψηφιακό τομέα και άρα τον εργαζόμενο εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και την αγορά εργασίας αυτή το, την ψηφιακή αγορά, ας πούμε. Δεν είναι σωστό να αφήσουμε στο ελαιό τους εργαζόμενους. Αυτά, κατά τα άλλα νομίζω η έκθεση αυτή είναι πολύ καλογραμμένη. Πρέπει να κάνουμε κάποιες επιμέρους βέβαια τροπολογίες, αλλά γενικά είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζωρίνιο είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή Ο ανταγωνισμό στο ψηφιακό τομέα είναι πολύ σημαντικός αν η Ευρώπη θέλει να παίξει ένα ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά στις προηγούμενες ψηφιακέ επαναστάσει, εμείς δεν τα καταφέραμε. Τώρα την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι τη νέα ψηφιακή αγορά να, τη να λάβει εκεί, να ληφθούν υπόψη νέε τεχνολογίε, Να μην ξεχνάτε ότι αυτέ οι νέε τεχνολογίε θα πρέπει να θέσουν εκ νέου την, ε, την Ευρώπη στην παγκόσμια αγορά, την ψηφιακή αγορά, χωρίς να αμφισβητήσουμε όμως τις αξίες, τα δικαιώματα και την προστασία του πολίτη. Θα πρέπει η γνωμοδότησή μας να είναι πιο σωστή. Στη γνωμοδότηση μιλάμε για τις υποδομές. Σήμερα ψηφίσαμε ένα τμήμα του κώδικα επενδύσεων που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό το στοιχείο για τα δίκτυα της πέμπτης γενιάς, γιατί ψηφίσαμε και την ε, γενική πρόσβαση στο ίντερνετ, με δωρεάν πρόσβαση, έτσι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. θέλουμε η αγορά να είναι ανοιχτή, να είναι ανταγωνιστική, να μην υπάρχουν αποκλεισμοί, Ο κύριος Κομπατσέφ έκανε διάφορες παρατηρήσεις, τις οποίες στηρίζω απόλυτα. Τώρα θέλω να κάνω μια επίκριση στην έκθεση. Είναι πολύ αμυντική για τις εμπορικές συμφωνίες, ας πούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα πάνω σε αυτές τις συμφωνίες. Να μην είμαστε μόνο αμυντικοί. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους κανόνες ανταγωνισμού, να βάλουμε σε αυτές τις εμπορικές συμφωνίες Και μια άλλη πτυχή. Θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα επιλογής, προστασία των ελευθεριών, ε, ελευθερία επιλογής. Όλα αυτά είναι στοιχεία της ψηφιακής μας ταυτότητας και είναι ε, τμήμα της, ψηφιακή της ψηφιακής ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν, ούτως ώστε να παίξουν προς όφελός μας. Θα πρέπει να λειτουργήσουν και να υπάρξουν στην δική μας αγορά, την ψηφιακή ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Ευχαριστώ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ο με τμήματάρχης στη Γενική Διεύθυνση Μπορείου, Ραλφ Πίνε, έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τη Γενική Γραμματεία προέρχομαι. Έχω όμως σχόλια από του εκπροσώπους τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου που δεν μπόρεσαν να παραστούν σήμερα. Θα σας τα διαβάσω εγώ λοιπόν. Καταρχάς, Εκ μέρου τη Επιτροπή, θα ήθελα να σα πω ότι η Επιτροπή καλωσορίζει αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση. Ε, είναι ισορροπημένο, καλό έγγραφο και μπορούμε να υποστηρίξουμε τα περισσότερα από τα σημεία που αναφέρει. Ε, συμμερίζεται τις τρεις αρχές η Κομισιόν, ε, επί των οποίων θα πρέπει να στηριχθεί η Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Οι εμπορικοί κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ε, πρόσβαση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, να δώσουν επίσης ωφέλη για Ευρωπαίους καταναλωτές και να σεβαστούν και να διασφαλίσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτά είναι οι βασικοί πυλώνες και για το, τη στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο. Ε, προσπαθούμε ε, σε όλα αυτά τα θέματα που αναφέρει η έκθεση να τα καταφέρουμε. Παράδειγμα, ε, υποβάλαμε και σχεδιάσαμε μια, ένα πλήρε ψηφιακό κεφάλαιο στι ε, διαπραγματεύσει με το Μεξικό και την Ινδονησία. Ε, και η πρόσφατη συμφωνία επί τη αρχή με την Ιαπωνία μπορεί να θεωρηθεί ένα καλό ορόσημο γιατί έχει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο που ανταποκρίνεται ε, στα περισσότερα στοιχεία τα οποία αναφέρει η έκθεση και τα καλύπτει. Ε, καταγράψαμε τις προτάσεις που κάνει το σχέδιο γνωμοδότησης και μπορούμε να υποστηρίξουμε τις περισσότερες, αλλά δεν θέλουμε να εστιάσουμε σε κάτι που μπορεί να επιτευχθεί περισσότερο μέσω των εμπορικών συμφωνιών. Κάποια από τα θέματα που, έχουν που αφορούν ε, τη σαφή φορολογία και τα... τους δασμούς μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω άλλων πρωτοβουλίων. Διάφορα... Διάφοροι βουλευτές μίλησαν το θέμα των ροών δεδομένων. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι είναι ένα τομέα αυτός όπου η... Ο εσωτερικό προβληματισμό τη Κομισιόν δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι σαφέ ότι η σωστή ισορροπία θα πρέπει να επιτευχθεί ανάμεσα στην προώθηση μιας φιλόδοξης ατζέντα στην καταπολέμηση της ε, ψηφιακής, του προστατευτικού... ψηφιακού προστατευτισμού, ε, να μην υπάρχουν ε, περιορισμού, περι... ανεπίτρεπτος και ανεπιθύμητο περιορισμό των δεδομένων, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα βασικά δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων. Η Κομισιόν εξετάζει ακόμα το πού θα βρει την ισορροπία ανάμεσα αυτά τα δύο θέματα. Ε, η Κομισιόν προσπαθεί να δει, περιμένει μάλλον τις τροπολογίες των Ευρωβουλευτών και ε, της Επιτροπής και των άλλων Επιτροπών και θα το συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα όταν θα έχουμε το κείμενο στην τελική του μορφή. Ευχαριστώ εκ μέρους Επιτροπής. Ο κύριος ε, Πουτικόφερ, εκ μέρους μάλλον τον κύριο Πουτικόφερ, ο συντονιστής ο κύριος Τούρμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η έκθεση του Ράινερ, καταλαβαίνω, ικανοποιεί τους και ηγητές με τις θέσεις που προβάλλει. Έχει δίκιο ο κύριος Ζωρίνιο. Ε, κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει περισσότερο η προστασία των πολιτών ως προς τα δεδομένα, αλλά και της ε, βιομηχανίας. Ξέρουμε ότι υπάρχει βιομηχανική κατασκοπία ακόμα και από φίλιες δυνάμεις. Και υπάρχει και πιο πρόσφατο θέμα που έχει ανακύψει που είναι η φορολόγηση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Θα συμβεί, είναι θετικό, ε, θα πρέπει να εξισορροπείται και από τις αρχές και τις αξίες μας. Ο κύριος Μπουτικόφερ προσβλέπει στη συνεργασία μαζί σας για τις συμβαστικές για να βγει μια καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 3η Οκτωβρίου 2017, αύριο δηλαδή, 6 ώρα το απόγευμα. Tomorrow, dear friends. Αύριο είπαμε. Έτσι για να καταλάβουμε τι 3η Οκτωβρίου, αύριο. Και θα ψηφίσει η Ήτρη στις 6 Νοεμβρίου. 6 Νοεμβρίου ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση. Uh, Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση. Η κυρία Μπιανκόσκα θα καταφτάσει σε 30 δεύτερα, το πολύ ένα λεπτό, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Και θα περάσουμε στο σημείο 10. Ο Σονούπο. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Ήτρε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Έχουμε έναν διαρθρωμένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε και δύο προτάσεις επιτάπητος, ένα πρόγραμμα για την βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας με ένα προπολογισμό των τάξης μετακοσίων εκατομμύριων ευρώ για διετή διάρκεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την πρόταση αυτού του προγράμματος. Η εταιρεία μας είναι η κυρία Γκροστέτ. Και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αυτό το ντοσιέ το γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα στην αρχή του 19. Είναι πολύ σημαντικό για μας λοιπόν. Το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα, η ανανεωμένη ε, βιομηχανική στατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χαιρετίζουμε και η οποία ακολουθεί το, την πρόσφατη απόφαση του ε, Κοινοβουλίου για την οικοδόμηση ενός, μιας φιλόδοξης στρατηγικής, βιομηχανικής στρατηγικής. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την στρατηγική πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας και σημαντική για ολόκληρο το Κοινοβούλιο, αλλά και για την βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύρια Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα εδώ. Αρχικά ε, θα ήταν μια συζήτηση για θέματα άμυνας και ιδιαίτερα για την πρόταση, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανική Ανάπτυξη στον τομέα τη άμυνα και χαίρομαι που βλέπω την εισηγήτρια, την ε, κυρία Γκροστέτ, του ισχυώδει ε, εισηγητέ και μέλη των διαφορών επιτροπών που θα συμμετέχουν σε αυτή την σημαντική πρωτοβουλία. Διότι σίγουρα δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να την συζητήσουμε εντελεχώς. Σας ευχαριστώ λοιπόν που με καλέσατε αλλά ε, με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα επίσης να σας παρουσιάσω εν συντομία ίσως, γιατί ίσως να έχουμε τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ανανεωμένη στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής που ξεκινήσαμε πριν από τρεις εβδομάδες, δύο εβδομάδες. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την βιομηχανική πολιτική και μετά στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθώ με το πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας. Όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την μεγέθυνση για να ε, εξυγχρονίσουμε την βιομηχανία του μέλλοντος και αυτός είναι ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους ε, έχουμε δουλέψει σε αυτή τη βιομηχανική στρατηγική, γιατί διασφαλίζεται ότι έχουμε μία βιομηχανία που είναι ευφυής, καινοτόμος και βιώσιμη. Γιατί η βιομηχανία μας είναι ε, στην κορυφή και θα πρέπει να την κρατήσουμε αυτούς τους καιρούς ε, τεχνολογικής ανάπτυξης, τεχνολογικής επανάστασης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία ηγείται σε όλους αυτούς τους τομείς να είναι ευφυής, καινοτόμος και βιώσιμη. Και βέβαια θέλουμε η βιομηχανία να έχει ε, σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, μια βιομηχανία που να επωφελείται της κλίμακας και της αποτελεσματικότητας ε, μιας ενιαίας αγοράς που λειτουργεί σωστά στην Ευρώπη και επίσης μια βιομηχανία που ε, ηγείται στον κόσμο προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξείδου του άνθρακου και μια κυκλική οικονομία. Αυτή η ανανεωμένη στρατηγική μας κτίζεται στη δουλειά που κάναμε στην, σε άλλες δράσει, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, την διαστημική στρατηγική. Η στρατηγική είναι βασισμένη σε έξι πυλώνες. Ε, δεν ξέρω αν θα έχουμε τον χρόνο σήμερα, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε αυτό, γιατί επεξεργαστήκαμε πολύ αυτό το θέμα. Μας πιέζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, η βιομηχανία και εσείς και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, να παρουσιάσουμε αυτό το έγγραφο. Στηρίζεται σε έξι πυλώνες, λοιπόν. Πρώτον, η ενιαία αγορά ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Και δεν σημαίνει ότι θέλουμε να καταρρύψουμε απλώς τους φραγμούς. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και νέες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Δεύτερον, θέλουμε να αναβαθμίσουμε την βιομηχανία για την ψηφιακή εποχή. Θέλουμε να έχουμε περισσότερη χρήση εμφυών τεχνολογιών σε, στην βιομηχανική αξιακή αλυσίδα, επίσης να περάσουμε σε μια οικονομία κυκλική με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου και εδώ ε, θέλουμε περισσότερες κεφαλογικές ε, επενδύσεις, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πέμπτον, στήριξη της καινοτομίας στη βιομηχανία. Για παράδειγμα, εδώ στηρίζουμε την χρήση και αξιοποίηση των ε, βασικών τεχνολογιών εφαρμογής και τέλος σε παγκόσμιο επίπεδο ανταγωνιζόμαστε. Ε, ξέρουμε ότι ε, το ανοιχτό εμπόριο βασισμένο σε κανόνες είναι απαραίτητο. Η αμοιβαιότητα, για παράδειγμα πρόσβαση στις αγορές προμηθειών, είναι κάτι το οποίο αναμένεται και είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε σε αυτό το έγγραφο. Ελπίζω ότι θα είστε διατεθειμένοι να το συζητήσουμε, ίσως όχι τώρα, αλλά ε, στο εγγύς μέλλον, για να μας στηρίξετε στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, διότι είναι, ελπίζω, ένα πολύ συνεκτικό έγγραφο που συνάδει με όλες τις προηγούμενες ε, πρωτοβουλίες μας. Τώρα, για το ε, πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας. Ε, ξεκινήσαμε το Ταμείο Άμυνας στις 7 Ιουνίου. Και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό στις προσπάθειες ανάπτυξης μιας ε, αμυντικής βιομηχανίας που μπορεί να έχει αποτελέσματα, να έχει τις δυνατότητες να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις ασφάλειας στην Ευρώπη. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, θα βελτιώσει τη συνεργασία σε όλους τους τομείς και σε ό, στον αμυντικό τομέα και σε όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό εδώ έχει, το έχω ήδη αναφέρει ότι έχει δύο πυλώνες, έρευνα και ικανότητες, δυνατότητες. Ο ερευνητικός πυλώνας ε, ήδη ε, έχει ξεκινήσει με το πιλωτικό έργο και την προπαρασκευαστική δράση με 90 εκατομμύρια ευρώ για διάρκεια τριών ετών. Έχει ξεκινήσει η πρόσκληση υποβολή ε, προσφορών για δύο συγκεκριμένα έργα, ένα μη ανδρομένο σύστημα και στρατιώτες για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή το συζητάμε για το πρόγραμμα εργασίας του 2018. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μέχρι τώρα στήριξή σας χωρίς ε, τη δράση σας, ιδιαίτερα ε, τη δράση του κυρίου Γκάλερ, ε, στην στήριξη της κατανομής του προϋπολογισμού η προπαρασκευαστική δράση δεν θα υπήρχε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και επίσης αυτό το μέρος θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, εξειδικευμένο πρόγραμμα έρευνας στον τομέα της άμυνας για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό το MFF. Θα ήθελα να συζητήσουμε όμως τον, τον πυλώνα των δυνατοτήτων, διότι αυτό αναφέρεται σε στοιχεία κλειδιά του προγράμματος της ε, βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας. Αυτή η Επιτροπή μαζί με τη ΣΕΤΕ, την ε, Επιτροπή Προεπολογισμού και την ΙΜΚΟ θα συζητήσουν τα θέματα αυτά στους επόμενους μήνες. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, που η Επιτροπή παρουσιάζει ένα τέτοιο πρόγραμμα για σκοπούς που σχετίζονται ε, με την άμυνα. Άρα είναι επαναστατικό, είναι κάτι που ίσως αλλάξει τα δεδομένα. Έχει δύο στόχους που ενισχύουν ο ένας τον άλλον. Πρώτον, στήριξη της ανταγωνιστικότητας ε, της βιομηχανίας της άμυνας και γι' αυτό επιλέξαμε τη νομική βάση ανταγωνιστικότητα ε, της βιομηχανίας, άρθρο 173 και δεύτερο στόχος είναι να επιτρέψει στην Ευρώπη προοδευτικά να ασφαλίσει τη δική της ασφάλεια και τη μη εξάρτηση. Αλλά το κάνουμε μέσα από την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα του τομέα της άμυνας. Και αυτό είναι ο κυριότερος σκοπό του προγράμματος και αυτό προτείνουμε να κάνουμε. Διότι οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. 80% των προμηθειών στην άμυνα γίνονται σε εθνικό επίπεδο, σε εθνική βάση και αυτό ε, οδηγεί σε επεκαλύψεις, σε μη αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα ε, υπάρχουν 178 οπλικά συστήματα στην Ευρώπη τις περισσότερες φορές δεν είναι ε, διαλειτουργικά. Σε σύγκριση υπάρχουν 30 στη ΣΥΠΑ τέτοια οπλικά συστήματα. Και υπάρχουν πολύ περισσότεροι τύποι ελικοπτέρων από κυβερνήσεις ε, που θα μπορούσαν να, αγοράσουν στην Ευρώπη, να τα αγοράσουν στην Ευρώπη. Σπαταλούμε πόρους, σπαταλούμε λεφτά και ε, υπολογίζεται από το Ευρωκοινοβούλιο το κόστος ε, της μη Ευρώπης στον αμυντικό τομέα υπολογίζεται στις 25 δις και 100 δις ετησίως. Ε, γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα ε, βιομηχανικής ανάπτυξης με χρηματοδότηση 500 εκατομμυρίων για τα τελευταία δύο χρόνια, το 19 και το 20. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να δώσουμε κίνητρα για συνεργασία, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συγχρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη των ε, αμυντικών δυνατοτήτων που θα συμφωνηθούν από τα κράτη-μέλη ως προτεραιότητες. Τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν πόν, λοιπόν ποιες είναι οι προτεραιότητες των δυνατοτήτων και η στόχη του προγράμματος, ε, μάλλον το πρόγραμμα στοχεύει μόνο ευρωπαϊκές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να, ε, να δυναμώσουμε τις δικές μας δυνατότητες και να κλείσουμε το τεχνολογικό χάσμα που υπάρχει με άλλα μέρη του κόσμου. Ε, θα καλυφθεί πρώτα η φάση του, των πρωτοτύπων, θα καλύψει και τις δοκιμές, το σχεδιασμό, την πιστοποίηση, τις μελέτες θα είναι υπομορφή επιδοτήσεων μέχρι 20% του συνολικού κόστους για τα, τα, πρωτότυπα και θα μπορούσε ε, να φτάσει μέχρι και 100% για άλλα, άλλες αναπτυξιακές δεδράσεις. Μπορεί να, ε, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στο 100% για άλλες αναπτυξιακές δράσεις. Για τα πρωτότυπα, για δυνατότητες 20-30%, αλλά μέχρι και 100% για άλλες δράσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν. Τι θέλουμε από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δεσμευτούν ε, να χρηματοδοτήσουν από κοινού την ανάπτυξη δυνατοτήτων, αλλά και να προμηθεύουν το τελικό προϊόν. Αυτό είναι ο τρόπος που κινητροδοτούμε τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε αυτό το τομέα. Δεν θα επικαλύψουμε ε, υπάρχοντα συστήματα, θα στηριχτούμε στις εξουσίες που μας ανατέθουν οι συνομοθέτες για την υλοποίηση της νομοθεσίας. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην ε, αναμίξουμε αυτό το πρόγραμμα με διακυβερνητικές διαδικασίες. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ ε, σύντομα σε δύο συγκεκριμένα σημεία τα οποία ξέρω ήδη συζητώνται είτε σε επίπεδο Συμβουλίου είτε στο Κοινοβούλιο. Πρώτον, το κατέστησα πολύ σαφές, το έχω ήδη πει και το επανέλαβα, ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι μόνο για τα μεγάλα τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη και για τις μεγάλες βιομηχανίες. Είναι ένα και προσπαθούμε να το σχεδιάσουμε να είναι ένα πρόγραμμα χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτό σε δικαιούχους από όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά φυσικά θέλω να είμαι πολύ σαφής, δεν θα επιβάλλουμε το geo-return ο στόχος, οι μας θα πρέπει να παραμείνουν ε, να παραμείνει στόχος η αποτελεσματικότητα βιομηχανική. Γι' αυτό προωθούμε τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από διαφορετικά κράτη-μέλη ε, για να ε, θεσπίσουν συμπράξεις, κονσόρτια στις αλυσίδες προμηθειών στον τομέα της άμυνας. Θέλουμε αυτό να ανοίξει τη διασυνοριακή συνεργασία. Γι' αυτό ε, προτείνουμε ότι το μερίδιο του προπολογισμού να ε, αφιερώνεται στις μικρομεσαίες. Η γεωγραφική ισορροπία επίσης θα εξαρτηθεί από τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα κράτη-μέλη. Ε, αυτό που αναζητούμε τώρα είναι αξιόπιστα διαφορετικά ε, έργα τα οποία μπορεί να προτείνουν τα κράτη-μέλη. Θα εξτάσουμε πολύ προσεκτικά τις προτάσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να φτιάξουμε τους κανόνες που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες μας, όχι μόνο στις μεγάλες βιομηχανίες και όχι μόνο στα μεγάλα κράτη-μέλη. Θα μια μεγάλη επιτυχία αυτό για το πρόγραμμα. Δεύτερον, στο 500 εκατομμύρια προπολογισμού θα ήθελα να εξηγήσω λίγο αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά το περιορισμένο χώρο ε, ελιγμών που έχουμε με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, ταυτόχρονα το ξέρουμε από την αρχή ότι αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, αν θέλουμε πραγματικά να ε, πετύχουμε ε, την ανταπόκριση των κρατών μελών στη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δεσμεύσουμε ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκά κονδύλια και ε, σημαντικά ποσά. Γιατί αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο ε, δίνει κίνητρα στην συνεργασία σε αυτό το τομέα. Και ε, παρόλο που από την αρχή είχαμε πλήρη στήριξη από όλα κράτη-μέλη, είναι κάτι αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τα κράτη-μέλη. Και το κάναμε πολύ προσεκτικά, αναμειγνώντας φρέσκα λεφτά, αν θέλετε, από τα περιθώρια και ανα, επαναδιαθέτοντας, θέτοντας από τα υφιστάμενα κονδύλια. Και θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι κανένα από τα τρέχοντα έργα δεν θα καθυστερήσει και ότι δεν θα επηρεαστεί η μελλοντική παράδοση των διαφόρων προγραμμάτων. Ήταν δύσκολο το έργο μας και πήρε χρόνο, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Θα πρέπει να βρούμε μια πραγματιστική λύση, μια ρεαλιστική λύση για να αξιοποιήσουμε αυτά τα δύο χρόνια που απομένουν το 19 και το 20 ως περίοδος δοκιμής για το μέλλον στο τομέα της άμυνας. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα και για το πρόγραμμα ανάπτυξης της ε, βιομηχανίας είναι σε πιλωτικό στάδιο. Θα μας βοηθήσουν και είναι γι' αυτό που ήθελα να το συζητήσω μαζί σας, διότι θα μας βοηθήσουν να ε, προσδιορίσουμε κατά πόσο οι, τρόποι και οι κανόνες είναι οι σωστοί για το μέλλον για το επόμενο MFF. Είναι επίσης μια δοκιμή των ικανοτήτων των δομών των ευρωπαϊκών θεσμών για να συζητούν, να διαπραγματεύονται και ευελπιστούμε ότι θα συμφωνήσουν και σε αυτά τα καινοτόμα προγράμματα που σχετίζονται με την άμυνα. Και σίγουρα δεν μπορούμε να αποτύχουμε σε αυτό το στόχο μας. Η Επιτροπή έχει προχωρήσει σε μια ανεπροηγουμένου σε αυτό το πρόγραμμα και να πω και το τώρα στους συνομοθέτες να ακολουθήσουν στο ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας και ξέρω υπάρχουν πολλά τεχνικά σημεία, τα ανέφερα ήδη. Ξέρω ότι μπορώ να στηριχθώ στη δική σας ε, ε, βοήθεια σε αυτή την Επιτροπή αλλά και στις άλλες ε, που προανέφερα και που σχετίζονται. Εάν θέλουμε το πρόγραμμα να είναι λειτουργικό, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, να είναι λειτουργικό από το 2019, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν εδώ την εισηγήτρια την κυρία Γκροστέτ που έδωσε αυτή την όθηση για ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά το timing. Αυτό είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε γιατί η Εστονική Προεδρία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια γενική προσέγγιση ήδη από τον Νοέμβριο, τον επόμενο μήνα. Και η συνεργασία με εσά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι θεμελιώδης, πολύ σημαντική. Μπορείτε να στηρίζετε στην πλήρη στήριξή μου και είμαι διαθέσιμη να απαντήσω σε ερωτήσεις. Στηρίζομαι στη βοήθειά σας και στο θέμα της βιομηχανικής στρατηγικής και στο θέμα του προγράμματος στον τομέα της άμυνας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για όλη αυτή την ενημέρωση και για τις τελευταίες προτάσεις σας. Πολύ συγκεκριμένες και ε, ε, δίνουν μια όθηση σε όλο αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχουμε εισηγήτρια και σκιώδες εισηγητές και ομιλητές αλλά και εκπροσώπους της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θέλω να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Ήτρε ότι η γενική ιδέα ενός τέτοιου προγραμματός είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για το βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης και ε, προέρχεται από την υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ. Εκείνοι ήταν οι εμπνευστέ. και σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι. Βεβαίως η βιομηχανική πολιτική είναι δική μας αρμοδιότητα, γι' αυτό το συζητούμε εδώ, αλλά εσείς ήσασταν οι ε, πατέρες της ιδέας αυτής και είστε πάντα πρόσδεκτοι. Ε, στην Ήτρε. Πάντα φυσικά σας δεχόμαστε με χαρά. Τώρα είναι απαραίτητη η ε, παρουσία σας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε εδώ. Η κυρία Σιγήτρια πρώτη λοιπόν και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ε, εκπρόσωποι της ΣΕΝΤΕ ή ο εκπρόσωπος που παρευρίσκεται και ετοιμάζει και τη γνωμοδότηση. Opinion on the, on the basis of rule είναι βάση του άρθρου 54 του κανονισμού μας όλα αυτά και πάρα πολύ σημαντική γνωμοδότηση ΣΕΝΤΕ ε, βάση του άρθρου 54. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκροστέτ και μετά στους υπολείπους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κυρίως ε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο Μπιενκόφσκα για την παρουσία της απόψε ενώπιον μας. Αυτό δείχνει πόσο προσιλωμένη είναι σε μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική γενικότερα. Αλλά θέλω να σταθώ ιδιαίτερα ε, και να εγκύψω στην ευρωπαϊκή ε, αμυντική βιομηχανική πολιτική. Είναι τεράστια τα ζητήματα και τα όσα διακυβεύονται. Τα ξέρουν οι συνάδελφοι, το διεθνέ πλαίσιο, θα τα πει συνάδελφου από τη ΣΕΝΤΕ, η πρόκληση τη καταπολέμηση τρομοκρατία, αστάθεια πολλών χωρών ε, του κόσμου, αλλά και επανέρχομαι στη βιομηχανία, έχουμε το διεθνή ανταγωνισμό, την ψηφιακή επανάσταση, που φέρνουν και επιφέρουν νέε απειλέ, αλλά και νέε ευκαιρίε παράλληλα. Άρα, ε, είμαστε αντιμέτωποι ε, και μπροστά μάλλον σε ένα βιομηχανικό πρόγραμμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο περίπλοκες είναι οι προκλήσεις, τα προβλήματα αλλά και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φορέα ισορροπίας παγκοσμίω. Βεβαίως ε, είναι πολλές οι ενισχύσεις στην αμυντική βιομηχανία, καινοτομία, έρευνα, ε, θέσεις εργασίας για όλους τους πολίτες. Ό,τι δίνουμε στην ε, άμυνα ε, είναι αλληλένδετο και αλληλεπιδρά και με την πολιτική, τη μη στρατιωτική βιομηχανία. Άρα και η αμυντική βιομηχανία μας θα πρέπει να είναι ενεργή, ανταγωνιστική ε, και ε, σφίζουσα. Αυτό που μας ενδιαφέρει, το είπατε και εσείς κύριε Επίτροπε, είναι να είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα με ε, απαιτήσει αριστεία που αυτό θα κάνει τη διαφορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχέση με άλλε βιομηχανίε. Η αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη συνεργάζεται σε διάφορα έργα, αλλά είναι συχνά ακριβή αυτή η συνεργασία και περιπλέκει τα πράγματα και τα προγράμματα. Άρα, ε, η πρόταση κανονισμού για ένα γνήσιο βιομηχανικό πρόγραμμα αποτελεί εξαιρετική βάση για να δώσουμε αυτή την όθηση που έλειπε μέχρι σήμερα στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Λοιπόν, κυρία Επίτροπε, αναφερθήκατε σε διάφορα προβλήματα και είναι γεγονός ότι όταν γίνεται λόγος για βιομηχανική, ε, πολιτική, αμυντική βιομηχανία, ε, είναι με βιομηχανική πολιτική αλλά και θέματα άμυνας και είναι πολύ ευαίσθητα αυτά γιατί είναι κατεξοχήν ε, ε, θέμα ε, κρατικής κυριαρχίας των κρατών μελών η άμυνα. Ε, οπότε, κύριε Επίτροπε, υπάρχουν κάποια σημεία που θα χρειαστεί να αποφασίσετε ή να αποφασίσουμε, γιατί δεν τα περιλαμβάνει η έκθεση. Και έχω ένα σημαντικό ερώτημα. Ποιο είναι ο προπολογισμό, έγινε λόγο για 500 εκατομμύρια για την επόμενη διετία, μάλλον 19-20 και για την επόμενη ε, δημοσιονομική προγραμματική περίοδο ακούμε μέχρι και 10 δισεκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά. Προφανώς το κοινοβούλιο μας και φαντάζομαι και οι πολίτες, οι συμπολίτες μας δεν θα κατανοούσαν το να μην δοθούν αυτά τα χρήματα ε, με άμεσο τρόπο σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εύκολα το λες αυτό, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο στην πραγματικότητα, γιατί ορισμένες ε, ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν συμφωνίες, συμπράξεις, κοινοπραξίες, μετοχές ε, και με εταιρείες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς θα συνταχθεί αυτό και πώς θα διαρθρωθεί έτσι ώστε να πιάνουν τόπο τα χρήματα αυτά και να καταλήγουν σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Προτείνατε αυτό το κανόνα του 50% των μετόχων να είναι σε ευρωπαϊκά χέρια, αλλά όπως κάθε κανόνας ε, είναι άκαμπτος. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε ένα κανόνα και να προσαρμόσουμε κάπως ε, αυτά που προτείνουμε έτσι ώστε να έχουμε τα έγκαιο ότι θα χρηματοδοτηθούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χωρίς να εμποδίζουμε τη δράση τους και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Επίσης, επιμείνατε στην ανάγκη να ε, εποφεληθούν από τη χρηματοδότηση αυτή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, συμφωνώ απολύτως. ακριβώς για να συμμετέχουν όλα τα κρατη και να προσιλωθούν σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει το κάθε κράτος να αισθάνεται ότι ε, το αφορά ε, αυτό το πρόγραμμα, με τι άλλο τις μικρομεσαίες του. Αλλά κυρία Επίτροπε θα πρέπει να παραμείνουμε ευέλικτοι ε, στο θέμα αυτό, διότι αν είμαστε υπερβολικά αυστηροί στην καθοδήγησή μας, δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουμε ε, τις αμυντικές βιομηχανίες από τη συμμετοχή. Τι θα μας προτείνατε λοιπόν για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πιο ακριβείς, σεβόμενοι πάντα την ευελιξία σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, our colleague, ε, Mr. Pascu. Ο κ. Πάσκου. Εκπροσωπεί την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ, την Άμυνας ασφαλείας και άμυνας. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στη σημαντική αυτή συνεδρίαση. Έχω... Έχω πέντε πράγματα που θέλω να θέσω. Καταρχάς, πρέπει να σπάσει μια ανθρωπία συγκεκριμένη. Η αμυντική βιομηχανία μέχρι τώρα ήταν εθνική υπόθεση. Γιατί η άμυνα ήταν εθνική υπόθεση. Μέσα σε αυτό το καλούπι δουλεύουμε. Οι βιομηχανίες μας εξαρτώνται από τις παραγγελίες των εθνικών κυβερνήσεων. Τώρα είμαστε αναγκασμένοι να βγούμε από αυτή τη λογική, από την οτροπία και να στραφούμε προς τη διεθνή αγορά, να, είμαστε, να έχουμε το βλέμμα πιο ανοιχτό. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε από αυτό το φραγμό, αυτή την οτροπία πρέπει να την ξεπεράσουμε. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες και υπάρχουν και παραδείγματα στη μελέτη που συνοδεύει μιλάμε, που συνοδεύει την πρόταση, μιλάμε για τη μελέτη του προσωπικού, όπου υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία και ξαφνικά 22 άλλα παρόμοια στοιχεία που προσπαθούν να ανταποκριθούν σε 22 μεμονωμένες ε, αιτήσει. Ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε το διάλογο να δούμε τα θέματα των απειλών και να τα καταλαβαίνουμε μονοσήμαντα. Είναι σημαντικό, είναι μια πολιτική διαδικασία. Αν θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των στοιχείων που παράγουμε, των μονάδων που παράγουμε, ας πούμε, στην αμυντική βιομηχανία, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Επίσης, αναπόφευκτα θα υπάρχουν και κάποια, μη, ε, κομμάτια που δεν φτιάχνονται στην Ευρώπη που εσωματώνται στο τελικό προϊόν μέχρι να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες να αντικαταστήσουν και μέχρι να, να το καταφέρουν αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ούτω ώστε να είμαστε σε θέση τελικά να έχουμε ένα προϊόν που λειτουργεί. Ακόμη και αν έχει κάποια κομμάτια, κάποια ανταλλακτικά, κάποια στοιχεία, πούμε, τα οποία δεν έχουν παραχθεί στην, στην Ευρώπη. Έτσι. Τέταρτον. Συνήθω. όταν οι χώρε αγοράζουν όπλα, από την Αμερική, α πούμε, δεν το κάνουν μόνο γιατί θέλουν αυτό το προϊόν. Το κάνουν βεβαίω και για την πολιτική εγγύηση που συνοδεύει το προϊόν. Επομένω, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίση να σκεφτεί και αυτή την πτυχή. Γιατί όταν λε, να, ένα καλό ευρωπαϊκό προϊόν, α πούμε. Ποιο θα έρθει να με υποστηρίξει όταν το χρειαστώ. Και εμεί τι λέμε, και 27 θα έρθουμε. Τι σημαίνει αυτό, κανένα βέβαια. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνεχίσουμε τη συνεργασία, ούτω ώστε να αυξήσουμε αυτή την αμοιβαία πολιτική στήριξη, αν θέλουμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα να είναι ελκυστικά τελικά. Τελευταίο σχόλιο, το οποίο αναφέρθηκε ήδη και χαίρομαι γι' αυτό. Όλοι θα πρέπει να έχουν κίνητρα να συμμετάσχουν. Δεν θα πρέπει να είναι ακόμα μία περίπτωση όπου οι μεγάλε εταιρείε πουλάνε στι χώρε τα προϊόντα του, α πούμε. Αυτό το καταλάβαν πολύ καλά στην Κομισιόν και χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιε διατάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πάσκου. σα ευχαριστώ που ήρθατε. Σα ευχαριστώ που εκφράσετε και την άποψη τη Υποεπιτροπή. Είναι πολύ σημαντική για μα. Γιατί υπάρχει μεικτή αρμοδιότητα για όλο το φάκελο αυτό. Επίσης, και όλες οι συγητές τώρα από την Επιτροπή Ήτρε, ο κύριος Πόχε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρώ αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας βασικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αναπτυσσόμαστε, παρόλα αυτά δεν έχουμε επαρκείς ε, δυνατότητες στις αμυντικές μας δυνάμεις. Υπάρχει αμοιβαία συμφωνία ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας. Αυτό θέλει και πολιτική βούληση, αλλά χρειάζεται και επαρκή χρηματοδότηση. Αυτό το πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό εργαλείο για να βελτιώσουμε το ευρωπαϊκό αμυντικό δυναμικό. Έχει έχει ένα μεγάλο δυναμικό, όχι μόνο για να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα αυτό, αλλά πιστεύω ότι και για τη συζητήση στην τελική τη μορφή θα πρέπει να σκεφτούμε και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες όπως το ΚΑΣ, ε, πρωτοβουλίες για την ΚΕΠΑ κτλ. Χαίρομαι που η Κομισιόν δίνει μεγάλη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ότι θα συμμετάσχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, το πρόγραμμα θα πρέπει μέχρι το τέλος της δημοσιονομικής περίοδου να δώσει ωφέλη. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να ξεκινήσει στις αρχές του 2019. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό ζητάει να γίνουν σημαντικά συγκεκριμένα βήματα για την ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Ήδη το 2012, το 2016 και το Κοινοβούλιο έχει επαναλάβει πλιστάκης ότι είναι διατεθειμένο να στηρίξει και σχετική νομοθεσία. Αυτός ο κανονισμός μιλάει για χρηματοδότηση από συγκεκριμένα κεφάλαια του προπολογισμού. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ε, γιατί ε, κάποιοι προπολογισμοί θα πρέπει να κοπούν για να πάνε τα λεφτά εκεί στο μέλλον θα υπάρξει, ελπίζω να υπάρξει και χωριστή συνεισφορά από τα κράτη-μέλη. Θα ήταν πολύ χρήσιμο κάτι τέτοιο. Η οικοδόμηση μια ενό κοινού αμυντικού δυναμικού ή δυνατοτήτων αυξάνει και την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και στην αποτελεσματικότητά της. Τώρα, έχω να κάνω τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η μία είναι λίγο προκλητική. Το σχέδιο δεν ξεκαθαρίζει αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε τη χρηματοδότηση του ορίζοντα 2020, Horizon 2020. Δηλαδή Και απέρριψε το να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του Horizon 2020 για αμυντικούς σκοπούς. Δεν λέει τίποτα για αυτό το θέμα η Κομισιόν. Τι, τι γνώμη έχετε εσεί. Αν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα λοιπόν το 2019, στου πρώτου μήνε του 2019, θα έχει προχωρήσει ο... σε μια περίοδο όπου το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ακόμα ε, μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι ότι κάποιε βρετανικέ εταιρείε θα συμμετάσχουν επίση στο πρόγραμμα. Γιατί η αμυντική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Όταν εκδοθούν ε, υπό το άρθρο 14 οι εφαρμοστικές πράξεις, η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει το, το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο πια να μην είναι πια μέλος για το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας του προγράμματος, το, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του προγράμματος. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το θέμα. Τρίτον, τι απόκριση είχατε από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την πιθανή αύξηση της συνδρομής τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα. Από τους σοσιαλιστές, ο κύριος Κρασνοντέμσκι. Συγγνώμη, ο κύριος Κρασνοντέμσκι από το ECR, όχι από τους σοσιαλιστές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όλοι μας στην αίθουσα αυτή Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Και φυσικά το προτινόμενο πρόγραμμα θα συνεισφέρει σε κάτι τέτοιο. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, Επίτροπε, το οποίο το ανέφεραν και διάφορες συνάδελφοι. Είπατε ότι θα πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή τη στιγμή κάποια από τη φρασιολογία του κειμένου ή κάποια διατύπωση που ελπίζω και χάρη στη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τροποποιηθεί, μπορεί να υποδηλώνει ότι έχουμε κάποιους φόβους σε ό,τι αφορά το, το σημείο αυτό, το κατά πόσον είναι ανοιχτό σε όλους. Ελπίζω το πρόγραμμα αυτό να μην έχει τις ίδιες αδυναμίες με το ορίζοντα 2020. όπου 500 ερευνητικές οργανώσεις, ε, οι πιο δραστήριες του, της Ευρώπης, έλαβαν το 80% του συνολικού προπολογισμού. Δηλαδή να μην υπάρχει συγκέντρωση του χρήματος ε, σε συγκεκριμένες βιομηχανίες. Γιατί αυτές οι ήδη ισχυρές βιομηχανίες μπορεί να ισχυθούν περαιτέρω με κάτι τέτοιο. Φυσικά υπάρχουν κάποιες δηλώσεις στο κείμενο, όπως π.χ. η απέτηση να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις εταιρείε σε μεμονωμένα project του προγράμματος, σε μεμονωμένα έργα. Θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποια άλλα κριτήρια ίσως. Ε, γεωγραφική ποικιλομορφία, ας πούμε. Γεωγραφική διαφοροποίηση. Όχι όλες από την ίδια χώρα ή την ίδια περιοχή. Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε επίση ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στου φόρους που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Επίση, κάνουμε λόγο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Σω θα έπρεπε να μιλάμε για εταιρείε που έχουν ε, χαμηλό κεφάλαιο. α πούμε μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείε. Και ένα άλλο θέμα. Είναι η διαφορετική συνεργασία με την ΠΕΣΚΟ. ΠΕΣΚΟ. Πρέπει να δούμε το θέμα της διαρθρωμένης μόνιμης συνεργασίας. Ξέρουμε ότι οι κανόνες της συνεργασίας ΠΕΣΚΟ δεν έχουν ακόμη ε, θεσπιστεί. Δεν ξέρουμε ποια κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να αλληλεξαρτήσουμε αυτές τις δύο πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίερινγκ είναι η επόμενη ομιλήτρια που αντικαθιστά τον κύριο Ρικέ, ο οποίος είναι σκιώδης ηγητής. Εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δυστυχώς κολλείται ο κύριος Ντομινίκ Ρικέ, δεν μπορεί να παρευρίσκεται σήμερα ε, για τη συζήτηση αυτή. Καταρχάς θέλουμε να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ταχεία κατάθεση αυτής της πρότασης ε, για ένα λεγόμενο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Είναι ακρογωνιαίος λήθος αυτός ο κανονισμός για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία και ολοκλήρωση. Ας είμαστε σαφείς για τους στόχους. Θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε την έρευνα, την ανάπτυξη, ε, τα πρωτότυπα ε, στην άμυνα με 500 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τα τέλη της παρούσης προγραμματικής περίοδου ε, με υποστήριξη ε, οικονομιών κλίμακα, συμμετοχή τουλάχιστον δύο κρατών μελών, εναρμόνιση των πολιτικών και ε, δημιουργία ενός αμυντικού ευρωπαϊκού βιομηχανικού κλάδου που να είναι παγκόσμιο ανταγωνιστικός. Και πολλές φορές ε, ουδέν κακόν γες καλό. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία του Brexit για να προχωρήσουμε από κοινού, να συνεργαστούμε για να καθορίσουμε τους κοινούς στόχους και τα μέσα μας. Η χρηματοδότηση των δυνατοτήτων μας είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσει η Ευρώπη να αναπτυχθεί και να συντονίσει διάφορα αμυντικά προγράμματα και όχι μόνο. Είναι και το πρώτο βήμα προς μια ε, πραγματική ηγεσία της Ευρώπης, βιομηχανική, με ε, καινοτομία στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας. Επίσης θα έχει και θετικό αντίκτυπο γενικότερα στην οικονομία μας, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, η αμυντική βιομηχανία έχει βοηθήσει να προχωρήσουν οι τηλεπικοινωνίες, η διαστημική έρευνα και ε, άλλα ε, θέματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται συντονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κράτη-μέλη και εξίσου σημαντικό είναι να έχουμε προγράμματα προτεραιότητας που είναι επιλέξιμα για την χρηματοδότηση με ομοφωνία από όλα τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Ρικέ έχει και δύο ερωτήσεις να σας υποβάλει. Όταν κοιτούμε τις πηγές χρηματοδότησης αυτού του ταμείου, 145 εκατομμύρια προέρχονται από τη διευκόλυνση συνδέονται στην Ευρώπη, ΣΕΦ. Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα. Μπορείτε να την αιτιολογήσετε αυτή τη χρηματοδότηση. Και δεύτερον, πώς βλέπετε τη μεικτή διαχείριση ε, κρατών μελών Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην πράξη πώς θα γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Το μικρόφωνο της ήταν πολύ κακό. Λοιπόν, επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Μπουτικόφερ, σκιώδης ηγητής εξ ονόματος των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για πραγματική καινοτομία, είναι νεοτερισμός αυτό που κατατίθεται σήμερα. Μπορεί να συμφωνώ με τα κίνητρα, αν τα καταλαβαίνω καλά, αλλά Αν έχω καταλάβει καλά, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κινητροδοτήσει τη συνεργασία. Αλλά διαφωνώ με την προσέγγιση και τη μέθοδο που επιλέγει. Έχουμε συζητήσει στρατηγικές για καλύτερη ε, χρηματοδότηση χρόνια ολόκληρα χωρίς να τα εφαρμόζουμε όλα αυτά που λέμε για το πώς να πιάνουν τόπο τα χρήματα. Ούτε καν δεν έχουμε επιβάλει την οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες η οποία τουλάχιστον 6, 8 ε, χρόνια συγγνώμη, ε, ισχύει. Τώρα μας λένε ότι αν πάρουμε χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τα μοιραστούμε με τα κράτη-μέλη, ε, θα έρθει η ρηξικέλευθη λύση. Αμφιβάλλω όταν ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Οργανισμός για να προωθηθούν οι κοινέ προμήθειες, το ίδιο μας, παραμύθι μας είπανε, αλλά δεν έγινε πραγματικότητα. Νομίζω η πραγματική τομή θα έρθει μόνο αν τα κράτη-μέλη πιστούν ότι θα πρέπει να συνεργάζονται, αντί να συνεργάζονται μόνο στη χρηματοδότηση ή εφόσον υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουν τα χρήματα κατά τα άλλα 250 εκατομμύρια ε, ετησίως για δύο χρόνια, ε, δεν θα φέρουν και την τεράστια αλλαγή. Και αν κοιτάξουμε ε, και τα ειδικότερα στοιχεία, αυξάνονται οι αμφιβολίες Ένα πρόγραμμα που θα απαντά σε όλα τα κριτήρια θα είναι τόσο άριστο και εξαιρετικό, οπότε γιατί να χρειάζεται επιπλέον ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να απογειωθεί. Πετάει και μόνο του. Η ανταγωνιστικότητα είναι μια πρόφαση δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω. Τα ξέρουν οι πάντες αυτά. Χρησιμοποιείται διότι υποτίθεται ότι θα δώσει νομική βάση στα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι επειδή χρειαζόμαστε πραγματικά ευρωπαϊκά κονδύλια για το σκοπό αυτό, για να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα από τη μια πουλάμε περισσότερα όπλα από όσα θα έπρεπε σε όλο τον κόσμο και από την άλλη αν μειώσουμε τις δαπάνες τότε θα βοηθήσουμε την ανταγωνιστικότητα γιατί υπερδαπανούμε έτσι ώστε να ανθούν εις βάρος των χρημάτων των φορολογουμένων ακόμα και εταιρείε που δεν είναι κερδοφόρες. Άρα αν θέλουμε να προάγουμε την ανταγωνιστικότητα δεν αυξάνουμε τη δική μας χρηματοδότηση. Επίσης πώς να το πω τώρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανητική η πρόταση που λέει ότι θα πάρετε λεφτά από το ΣΕΦ για να τα δώσετε εκεί. Μα είμαστε σοβαροί για το οικονομικό και βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε την αμυντική βιομηχανία παίρνοντας χρήματα από το Connecting Europe. Συν από το πρόγραμμα προήγησης με δορυφόρο αυτό είναι προπετούμενο για καλή αμυντική συνεργασία αυτό το πρόγραμμα. Γιατί να παίρνουμε χρήματα από τη μια τσέπη να τα βάζουμε στην άλλη. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Νομίζω θα πρέπει να αλλάξουμε τακτική και προσέγγιση και να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν. Είναι σωστό αυτό. Να κάνουν κοινά μαζί, ε, αλλά ο δρόμος δεν είναι να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία ε, να επικρατήσει εδώ το αμυντικό λόμπι. Ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ τώρα ο κύριος Ηλικιώτης, επόμενος και Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πρώτα πρώτα να πω κυρία Επίτροπη Πιγκόφσκα, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Ε, παρουσιάσετε πρώτα τη βιομηχανική πολιτική και μετά το νέο αμυντικό σχέδιο και την αμυντική βιομηχανία που κατά την άποψή μας με τον τρόπο που προωθείτε, ακυρώνει ε, το νέο αμυντικό σχέδιο την όποια προσπάθεια για στήριξη της βιομηχανίας. Ε, εμείς διαφαινούμε κάθετα, όχι μόνο διαδικαστικά, διότι αυτό το νέο αμυντικό σχέδιο εξαγγέλει κατά την άποψή μας την απαρχή της διαδικασίας για πλήρη στρατιωτικοποίηση της Ένωσης. ζητείτε δηλαδή να γίνουν επενδύσει στον τομέα της άμυνας, να ενισχυθεί η στρατιωτική βιομηχανία, ώστε να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ισχυρότερο εταίρο στο στρατιωτικό τομέα. Προτείνεται δηλαδή η δημιουργία μόνιμου στρατιωτικού δομών, ενό Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Άμυνα, με προπολογισμό 38,5 δισεκατομμύρια παρακαλώ, από το 20 μέχρι το 2027. Δηλαδή 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού, για ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και για πρόθεση της έρευνας για στρατιωτικούς σκοπούς. Όλα αυτά κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι είναι οι πραγματικές ανάγκες σήμερα της οικονομίας των λαών και ε, των κοινωνιών στην Ευρώπη. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα κονδύλια αφαιρούνται ήδη από συγκεκριμένα αναπτυξιακά προγράμματα, αναφέρθηκε ε, και από τον προλαλήσαντα μερικά από αυτά τα στοιχεία. Αφού υπάρχει διαθέσιμο ένα τόσο μεγάλο κονδύλι, γιατί δεν το αξιοποιείτε για την πρόθεση της επαναβιομηχανοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρξει ξανά κοινωνική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον Νότο που έχει πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και τι νεοφιλεύθερε πολιτικέ ιδιότητε. Γιατί δεν χρησιμοποιείται το διαθέσιμο κονδύλι για να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιομηχανία, με άξονα την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, όπω αναφέρατε και στην εισαγωγική σα παρέμβαση, επιτυχάνοντα τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασία και πρόθεση μια ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας και όχι ε, στρατιωτική ε, βιομηχανία και έρευνα προς όφελος κυρίως των πολυεθνικών δυνάμεων, των πολυεθνικών εταιριών. Οι προτάσεις που προωθούνται για δυναμητική βιομηχανία όχι μόνο δεν θα αφαιρέσουν την όνωση, αλλά κατά την άποψή μα θα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για τους λαούς. Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι πολίτες που σε μεγάλα τμήματα φτωχοποιούνται είναι αναπτυξιακές πολιτικές για όθηση της πραγματικής οικονομίας, για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας. Δεν θέλουμε κονδύλια για πολέμους. Γιατί στήριξη αμυντικής βιομηχανίας αυτό σημαίνει. Σημαίνει ενίσχυση της επεμβατικής πολιτικής σε πολλές περιοχές που σήμερα υπάρχουν πολέμους. Εμείς αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει πρωτοβουλίες για πλήρη αποστρατιοποίηση, για πρόθεση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για επαναβιομηχανοποίηση της Ένωσης και για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της κοινωνίας και όχι οι ανάγκες της πολεμικής βιομηχανίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για Έκλεισε ο κατάλογο τελείωσε αυτός ο κατάλογος των σχεδόν εισηγητών και των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Τώρα θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπου ομιλητέ, στου υπόλοιπου βουλευτέ, ο κ. Σαλίνη πρώτος. Ευχαριστώ. Το πολύ δύο λεφτά παρακαλώ συνάδελφε, γιατί έχουμε ένα τεράστιο κατάλογο. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις, πολύ σύντομες θέλω να κάνω. Πρώτον, για την δομή των προτεραιοτήτων ε, γύρω από τις οποίες ε, διαρθρώνεται αυτό το πρόγραμμα. Θα είμαι σύντομο, γιατί τα βασικά στοιχεία υπόθηκαν από την κυρία Γκοστέτ. Στο άρθρο 7 η πρόταση αναφέρεται στο σε ό,τι αφορά το ownership στο 50%. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μα κατά την απόψή μου, ε, στι προτεραιότητε του προγράμματο. Και η προτεραιότητα του προγράμματο είναι από τη μία να έχει πολιτικό χαρακτήρα η άμυνα, η αμυντική βιομηχανία συνδέεται καταρχάς με την νέα πολιτική για την άμυνα. Επομένως, βασικό είναι να έχουμε μια βασική και στεναρή αμυντική πολιτική και μέσω αυτής οι χώρες καθορίζουν το, το δυναμικό και τις προτεραιότητες. Και το δεύτερο θέμα είναι το βιομηχανικό, το καθαρά βιομηχανικό. Το 50% του ownership είναι μία ε, άκαμπτη πρόβλεψη. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η κυρία Γκροστέτ. Το σωστό θα ήταν ε, να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δηλαδή θα πρέπει το, να θέσουμε να λάβουμε υπόψη μας το know-how στην Ευρώπη και να, την Ευρώπη να την κάνουμε κέντρο του know-how. Ε, το κέντρο της άμυνας να γίνεται στην Ευρώπη και όχι αλλού. Πέρα από το ownership, πέρα από το ποιο είναι ο ιδιοκτήτης. Τουλάχιστον να μην κολλάμε εκεί. ούτω ώστε τα θετικά, ας πούμε, ε, στοιχεία ε, και σε πολιτικό επίπεδο και σε βιομηχανικό επίπεδο να τα, να, να τα ε, καρπούμεθα εμείς. Επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας ε, καίει αυτό το θέμα, αλλά τι εννοούμε εδώ πέρα. Οι διάφορες χώρες έχουν διαφορετικούς ορισμούς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε με πονηρό τρόπο και δόλιο τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι. Προσοχή λοιπόν, προσοχή. Και δεν κάνω άλλες παρατηρήσεις. Περιορίζομαι σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαλήνη. Ο επόμενος ομιλητής. κύριος Μαχτά. Ευχαριστώ. Ε, εγώ δεν θα πάρω πάνω από δύο λεπτά, αλλά σας παρακαλώ. Θα Α, μπορεί να, να χρειάζεται περισσότερο από δύο λεπτά, αλλά σας παρακαλώ την επίοικιά σας ε, για την αμυντική πολιτική. Μια ανανεωμένη στρατηγική, λέτε, για την αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Θέλω να μιλήσω πρώτα για τα θέματα και τα διακυβεύματα εκτός της Ένωσης και μετά για εντός της Ένωσης. Αλλά τα δύο είναι αλληλένετα. Θα το καταλάβετε. Και ε, το είπατε κι εσείς. Πώς θα οικοδομήσουμε μια βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χρειάζεται πρώτα απ' όλα πολιτική βούληση. Ε, την έχουμε, τη διαθέτουμε, την πολιτική βούληση, γιατί εδώ και 40 χρόνια η βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης και των κρατών μελών, γιατί και τα κρατημέλη κάνουν βιομηχανική πολιτική και έχουν ευθύνε. Ε, συνίστατο στο να πουλήσουν ε, τις εθνικές βιομηχανίες, να τις ιδιωτικοποιήσουν. Βλέπετε πρόσφατα στη χώρα μου είναι δύο τα μεγάλα θέματα και όχι μόνο ε, η υπόθεση Siemens Alstom που αγοράζει και η Φιγκαντιέρη που αγοράζει τα STX, τα ναυπηγεία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι οι συγχωνεύσεις εξαγορές σημαίνουν βιομηχανική πολιτική. Και ποια είναι η πραγματικότητα πώς η Ευρώπη θα αποκτήσει εκείνα τα εργαλεία, τα θεσμικά και τα πολιτικά για να καταπολεμήσει τα μαστόδων που είναι οι Κινέζοι, ε, Ινδοί και Αμερικανοί. Ε, τα θηρία, τα μεγαθύρια. Ε, είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένα όλα αυτά και πάρα πολύ στεγανοποιημένα. Αυτός ο ευρωπαϊκός πρωταθλητής ε, είναι εκ των όνων για να υπάρχουμε στην παγκόσμια αγορά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει δύο εταιρείες που συνεργάζονται. Είναι μια εταιρεία που τρώει την ε, μικρότερη. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν στην Ευρώπη είναι μια νέα πολιτική που να επανακαθορίζει τους κανόνες του ανταγωνισμού. Κύριε Πρόεδρε, λίγο την επίκαια είμαι και είναι σημαντικό. Δεν κάθομαι μέχρι τις 9.30 ώρα για να μιλήσω δύο λεπτά. Μα είπατε ότι θα μιλήσετε λιγότερο από δύο λεπτά. Το αντίθετο είπα, αλλά... Αν έχουμε χρόνο στο τέλος θα σας ξαναδώσω το λόγο. Αν θέλετε να μιλήσετε περισσότερο. Θα σας δώσουμε το λόγο στο τέλος, αν περισσέψει χρόνος. 30 ε, δεύτερα, να πω δύο φράσεις. Για κάθε φορά ε, το ίδιο έργο βλέπω. Ε, γιατί θα καταλήξω να πιστεύω ότι είστε θυμωμένος μας. Έλεγα λοιπόν, ότι το είπαμε και το επαναλάβαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ως αναφορά την παγκόσμια αγορά. Ακριβώς για να δει πού θα τοποθετηθεί εκεί και αν είναι οι ε, θέσεις μας δεσπόζουσες ή όχι. Ε, κοιτάξτε τι γίνεται στο αλουμίνιο στην Κίνα, τι γίνεται ε, στο σιδηρόδρομο στην Κίνα. Και μια που μιλάτε για τις ευθύνες των κρατών, ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε για μια βιομηχανική πολιτική που θα βάλει στα ευρωπαϊκά σύνορα ένα φόρο για το διοξίδιο του άνθρακα. Δεν σας θυμίζει τίποτα, Πρόεδρε. Ήταν στην έκθεσή είμαστε στο κείμενο και το βγάλανε. Και τελειώνω, τελειώνω εδώ. Τα κράτη-μέλη, λοιπόν, είναι πρόθυμα να σας παρακολουθήσουν. Ενώ τα ε, εργαλεία αμυντικά τα αμυντικά εργαλεία για το εμπόριο έχουν μπλοκαριστεί εδώ και τρία χρόνια. Ο κύριος Γκάλερ που εκπροσωπεί την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε, το έχω πει επανειλημμένα Κυρία Επίτροπε, είμαστε ευγνώμονε για την εξαιρετική δουλειά για την άμυνα που έχετε κάνει μέχρι τώρα και εσεί και ο Αντιπρόεδρο Κατάινεν και η κυρία Μογκερίνη έχετε επιδείξει ένα πραγματικό πολιτικό θάρρο και όσο και όραμα ε, καταθέτοντα ε, την ανακοίνωσή σα και την νομοθετική πρόταση κτλ και το έγγραφο ε, προβληματισμού για την άμυνα. Εμείς στο Κοινοβούλιο θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας ε, στο συγκεκριμένο τομέα. Συνάδελφοι, ήταν εξαιρετική η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσθέσει το πρόγραμμα αυτό που κυρίως χρηματοδοτούν τα κράτη-μέλη. Εμείς το ζητήσαμε από το Κοινοβούλιο για να έχουμε ε, περισσότερη προσήλωση και οικονομικές υποσχέσεις από τα κράτη-μέλη η διάδραση μεταξύ έρευνας και ανάπτυξης ε, μπορεί να μας εγγυηθεί ότι η κοινοτική χρηματοδότηση θα απορροφηθεί από τα κράτη-μέλη ε, στα διάφορα προγράμματα προμηθειών τα κράτη-μέλη χρειάζονται αμυντική συνεργασία για να έχουν καλύτερο εξοπλισμό. Ας πούμε, οι ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται ένα ευρωπαϊκό ντρόουν παρατήρησης, ε, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Ε, ορίστε, ε, θέλω να προτείνω κάτι, Επίτροπε, και να μοιραστώ μαζί σας μια ανησυχία. Έχουμε κάποιους συναδέλφους που αμφισβητούν γενικά ε, την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αμυντικά, αλλά και σε αυτό συμφωνώ με αυτό που προτείνεται. Το 173 ε, άρθρο να είναι η νομική βάση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά κυρία Επίτροπε, σε αυτή τη νομική βάση θα θέλατε να προσθέσετε μια ευρύτερη πολιτική βάση αναφερόμενη στο άρθρο 2.4 στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσετε ότι έχει αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα αμυντικά για να απαντήσουμε στους επικριτές και να δώσουμε περισσότερη νομιμοποίηση σε αυτή τη νομοθετική προσπάθεια. Και παραθέτω το εν λόγω άρθρο όπου αναφέρεται μια κοινή αμυντική πολιτική και στο 2.5 λέει σε κάποιους τομείς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αρμοδιότητες για εκτέλεση δράσεων ε, υποστηρικτική, ε, συντονιστική ή συμπληρωματική προ τι ε, δραστηριότητε των κρατών μελών που είναι αρμόδια για την άμυνα, αλλά εμεί έχουμε αρμοδιότητα να τα υποστηρίζουμε. Εκτός από το 173 να βάλουμε και το 2.4 και το 2.5 της ΣΛΕΕ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόγια, αντιπρόεδρος μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ουσιαστικά θα μιλήσω για την αμυντική βιομηχανική πολιτική, γιατί τα άλλα τα είπαν άλλοι συνάδελφοι. Πολύ λίγα πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο και γιατί τελικά η βιομηχανική πολιτική επιτέλους είναι μέσα στις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρώτο που έχω να πω είναι το εξής. θα πρέπει να, δούμε ποιες είναι οι θέσεις μας. Μέχρι τώρα είχαμε περιοριστεί στο να λέμε ότι η βιομηχανική πολιτική συμπεριλαμβάνεται στις επιμέρους πολιτικής. Σήμερα υπάρχει μια ουσιαστική βιομηχανική πολιτική που δίνει ε, την κατεύθυνση και σε άλλες πολιτικές όπως η εμπορική και άλλες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη βιομηχανική. Ε, άλλος στόχος. Σήμερα βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει κάποιους μεγάλους πρωταθλητές που θα πρέπει να βοηθήσουμε να είναι διεθνώς ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να ξαναδούμε το δίκαιο του ανταγωνισμού που γεννήθηκε όταν ο ανταγωνισμός ήταν εσωτερικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης έχουμε ένα πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα πρέπει να ε, υποστηριχθούν. Σήμερα δημιουργείται θέμενη αξία και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι εταιρείες όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Θα πρέπει να τις βοηθήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό εύκολο δεν είναι αλλά ξέρετε ότι έχουμε μικρομεσαίες που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας ε, στις χώρες μας. Να έχουμε καινοτόμα συστήματα και fast track ας πούμε εργαλεία για να ενισχυθούν όλα αυτά για την καινοτομία και την ολοκλήρωση. Και σε περιφερειακό επίπεδο και σε διακλαδικό. Επίσης θα πρέπει να ε, προωθήσουμε αυτή τη ψηφιακή επανάσταση που συνδέεται με τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες. Τώρα μιλούμε για επιχειρήσεις 4.0, είναι ψηφιακή εποχή. Έχει τελειώσει το παλιό το εργοστάσιο, η κατασκευαστική βιομηχανία στην Ευρώπη. Ε, έχουμε νέα δεδομένα, νέες αλλαγές, έχουμε ε, πληροφορίες, κατάρτιση σε κάποια κράτη-μέλη πραγματικά καταρτίζονται οι διεργαζόμενοι προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, είναι όλα αυτά τα στοιχεία σημαντικά ε, και θα πρέπει αυτή η ιδέα να βρει το δρόμο της και μέχρι την πολιτική. Σταματώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω μόνο το εξή ότι περιμένουμε ένα σχέδιο δράσης που να είναι ουσιαστικά δράση. Πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και επιχειρήσεις. Ο μιλητής επίσης εκπροσωπεί την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ, ο κύριος Ρίτς. Λίτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε στα Πολωνικά ο κύριος Λίτς. Ε, ήθελα να σας πω ότι εγώ είμαι Ευρωπαίος Σοσιαλδημοκράτης. που είναι υπέρ ενό ευρωπαϊκού στρατού, ευρωστρατού και pooling and sharing, δηλαδή συνένωση των δυνατοτήτων και κοινή χρήση και πολλά πράγματα τα βλέπω τελείως διαφορετικά από ό,τι ακούμε εδώ. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσουμε. Ε, χρησιμοποιείται εδώ ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, αλλά τα κράτη-μέλη ε, αποφασίζουν εκείνα για τις εξαγωγές τους, παραμένουν εθνικές. Έχουμε εγκρίνει τώρα μόλις μια έκθεση για μια ε, οδηγία για τις εξαγωγές και χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο κατάλογο εξαγωγών και δεν γίνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην συναποφασίζει και συνομοθετεί. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν την καινοτομία, το pooling και sharing, δηλαδή τις κοινέ δυνατότητες που θα χρησιμοποιούν από κοινού. Κάποτε τα είχε πει αυτά ο κύριος Γιούγκερ, αλλά τι γίνεται με την μετατροπή. Κάνετε μετατροπή της δουλειά σας για αυτά ε, για αυτές τις επιχειρήσεις που θα πρέπει να αλλάξουν ε, την παραγωγή τους γιατί ας πούμε από τα 15, τους 15 τύπους αρμάτων μάχης που έχουμε θέλετε να έχουμε μόνο δύο και τους υπόλοιπους 13 θα τους κάνουμε σε τι θα μετατραπούν, θα μετασχηματιστούν αυτές οι εταιρείε και οι βιομηχανίες γι' αυτό λοιπόν ζητώ να ε, πάτε προς τη σύγκληση και τα κράτη-μέλη να προωθήσουν το pooling και sharing με κοινοβουλευτική συναπόφαση η οποία απολύτως απουσιάζει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ως Ευρωβουλευτής θα πρέπει να εγκρίνω ένα προϋπολογισμό που θα συνεχίζει να περιστέλει τις δικές μου ελευθερίες και δυνατότητες συναπόφασης. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Στη συνέχεια τώρα ο κύριος Γκάιαρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ωραία που παίρνω το λόγο μετά το συνάδελφο Λίτς, γιατί μπορώ να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε εκείνος. Δεν ξέρω τι να θαυμάσω περισσότερο και τι να απορρίσω περισσότερο ακούγοντας την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τη συζήτηση εδώ. Αν απορρίσω περισσότερο για την πρόταση ή για τη συζήτηση εδώ διαφόρων επιτροπών. Είναι πολλά τα θαυμαστά που μας υπόσχεται αυτό το ταμείο που είναι και μικρός ο προπολογισμό. Μα τι ελαφρότητα είναι αυτή και επιπολαιότητα. Ε, αναφερόμαστε σε αριθμούς για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ήδη μας πονάνε τα 500 εκατομμύρια να τα βρούμε από τώρα. Μιλάμε για τα επόμενα. Ο συνάδελφος Μπιτικόφερ πολύ σωστά τα είπε. Η αντίσταση που θα έρθει όχι μόνο από την Επιτροπή Προπολογισμών από αλλού θα είναι μεγάλη. Και ένα τρίτο που με εκπλήσει και πραγματικά με έχει αφήσει άναυδο είναι αυτή η ανεμελιά για τα οικονομικά. Κυρίες και κύριοι, με το Brexit θα χάσουμε το δεύτερο μεγαλύτερο καθαρό συνεισφορέα. Από το Κοινοβούλιο δεν άκουσα ούτε μία πρόταση, ούτε μία εθνική αντιπροσωπή, ούτε μία ε, επιτροπή να λέει ότι υπάρχει η τάδε γραμμή του προπολογισμού και μπορούμε να δώσουμε χρήματα, α, καμιά ε, εκατοστή εκατομμυριάκια την περιφερειακή πολιτική, τη γεωργική πολιτική να τα δώσουμε στην άμυνα. Μα κάθε χρόνο ζούμε τα ίδια στη συζήτηση για τον προπολογισμό. Ακούω από το Συμβούλιο πάντα ότι θέλουμε να έχουμε αποθεματικό για πρόβλεπτα και αντιδράσεις κτλ. Μα αν μπορούμε να ανατρέξουμε στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να χρηματοδοτήσουμε κάτι, για να προάγουμε κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει. Και ακούω από την Επίτροπο ότι τα κράτη-μέλη περίμεναν να έρθουν πολλά κονδύλια. Εδώ δεν συζητάμε πια για χρηστή διαχείριση του προπολογισμού, για οικονομίες κτλ. Ε, στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός, αυξάνονται όμως οι προτεραιότητες. Ανησυχώ πάρα πολύ γιατί πολλά από τα τμήματα αυτού του προγράμματος θα τα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη διακυβερνητικά, θα περιορίσουν και θα περιστύλουν την ε, δημοκρατική έκφραση του Κοινοβουλίου και στην επιλογή ε, των προγραμμάτων τα κριτήρια δεν θα είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν και τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά ε, αυτά που συμφέρουν, συμφέρουν την αμυντική βιομηχανία κάθε κράτος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόιζινγκ. Και πάλι από την Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τους δύο προλαλήσαντες απολύτως. Πιστεύω ότι οι πολίτες στην Ευρώπη, άνδρες και γυναίκες, θα πρέπει να ενημερώνονται ανοιχτά και ειλικρινά περί πόσων δισεκατομμυρίων πρόκειται, πού θα βρούμε τα λεφτά και πόσα λεφτά θα δώσουμε ε, και από πού θα τα κόψουμε στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, ε, δεν μπαίνω στην ουσία. Και εγώ έχω μείνει άναυδη ε, για τον τρόπο με τον οποίο διαστρεβλώνονται τα πράγματα. Στη Γερμανία υπήρχε μια ταινία που έλεγε ότι δεν μας ταιριάζει, τον κάνουμε να μας ταιριάζει διαστρεβλώνουμε τα πράγματα. Ε, αμυντικές δυνατότητες, στρατηγική άμυνα, στρατιώτης του μέλλοντος και πράσινα άλογα. Ε, ουσιαστικά, αυτά έρχονται στην Επιτροπή Ήτρε. Και ε, έτσι παρακάμπτεται η απαγόρευση χρηματοδότησης που λέει το άρθρο 41.2. Το 2016 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί και παραθέτω για αντίστοιχο δείχνει ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα σε περίπτωση που έχει διπλό στόχο ή δύο στοιχεία ε, τότε υπάρχει το ένα το οποίο κυριαρχεί και το δεύτερο είναι δευτερεύον υποδέστερο. Δηλαδή ένα νομοθέτημα οφείλει να βασίζεται και να εδράζεται σε μία και μόνο νομική βάση και αυτό είναι το κυρίαρχο και τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Κατά την άποψή μου λοιπόν ε, είναι η ασφάλεια και άμυνα το βασικό και το ουσιαστικό και μέχρι στιγμής ο κύριος Μακάλιστερ και η κυρία Φωτίγκα, πρόεδροι των Επιτροπών ΑΦΕΤ και ΑΦΚΟ συμφώνησαν και ε, με παραπομπή αυτών των αρμοδιοτήτων προσπάθηκαν σαν να ε, το δώσουν στη ΣΕΝΤΕ και στην ΑΦΕΤ αυτό το θέμα και όχι στην Ήτρε. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Πώς επηρεάζει η νομολογία Ε, πώς επηρέαζε αυτή η νομολογία 263 του 2014, απόφαση 14 έκτου του 16 για το 137. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Κόχλιτσεκ, πρόεδρος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Άκουσα κάτι βλακίες εδώ πέρα ότι ενισχύοντας την αμυντική βιομηχανία μπορούμε να προστατευτούμε, να από τους τρομοκράτες. Αυτά είναι τώρα σαν χλαμάρες. Ας τα ξεχάσουμε, έτσι. Επίσης, άκουσα και κάτι άλλο. Ότι έχουμε 175 διαφορετικά ε, οπλικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να τα ενοποιήσουμε, δεν θέλουμε κάποιο ειδικό νομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ των κατασκευαστών. Και η υποστήριξη επίση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ηλίθιο. Οι μεγάλε επιχειρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δραστηριοποιούνται στην τομέα τη άμυνα. Αν θέλετε να βοηθήσετε την βιομηχανία, μην πάρετε πόρου από το ΣΕΦ ή από το ΣΑΤΝΑΒ. Να τα κρατήσετε εκεί τα λεφτά, στο Connecting Europe Facility, γιατί έτσι θα αναπτυχθεί η Ευρώπη. Ψάξτε αλλού να βρείτε πόρους. Γιατί αν αποφασίσετε να πάρετε από αυτά τα προγράμματα κονδύλια, στην πραγματικότητα κόβετε λεφτά και θέσει απασχόληση από αυτή την βιομηχανία. Από κάποιες βιομηχανίε, μάλλον. Και επίσης αν θέλετε να, προχωρήσετε, να στηρίξετε τη βιομηχανία, α κάνουμε ένα πρόγραμμα για τα νέα υλικά. Τα μεταλλικά και τα μη μεταλλικά, καθώς και για τα ηλεκτρονικά υλικά. Γιατί σε όλα τα συστήματα που έχουμε είναι, εισάγουμε υλικά τέτοιου τύπου. Από πού εισάγουμε παρακαλώ, από την Ινδία, την Κίνα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. κλπ. Και φυσικά αυτές οι εταιρείε αυτές τις χώρες φυσικά τελικά επηρεάζουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Θαυμάσια έρχονται τα πράγματα. Με τη σειρά μιλάμε. Πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι εκπλήσωμαι για την αφέλεια και την ελαφρότητα με την οποία συζητάμε πράγματα που πριν από λίγα χρόνια θα τα θεωρούσαμε ε, ανήκουστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αδιανόητα. Πρόκειται για μια κούρσα εξοπλισμού, δεν είναι μια οποιαδήποτε βιομηχανική πολιτική είναι η χρηματοδότηση ε, ενός ε, ε, στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος... στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκή κονδύλια και τα παίρνετε από την Connected Europe, από την προστασία του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής... και από άλλα προγράμματα και ερευνητικά που θα είχαν νόημα για το σκοπό αυτό. Και δεν είπατε ούτε κουβέντα και πραγματικά εκνευρίζομαι για το τι θα γίνει με το Brexit. Αν κοιτάξουμε τα κονδύλια, και ότι θα χάσουμε ε, πολλούς πόρους. Πώς θα το αντισταθμίσετε, πώς θα το χειριστείτε. Μα πώς βγαίνει αυτός ο λογαριασμός. Θα πάρετε τα λεφτά από τη συνοχή. Το ρώτησε και άλλος συνάδελφος. Ή από τη γεωργία. Ή από την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα αυτό. Πώς δικαιολογείται μια τέτοια πρόθεση που μας παρουσιάζεται εδώ. Αν κοιτάξετε τι γίνεται στη Νότια Ευρώπη. Ναι, εκεί η βιομηχανική πολιτική χρειάζεται γιατί χρόνια ολόκληρα αποδομήθηκαν, αποβιομηχανίστηκαν ολόκληρα κομμάτια, περιφέρειες της Νότιας Ευρώπη. Εκεί χρειάζεται επενδύσεις για τις υποδομές, στοχευμένα προγράμματα καινοτομία για τη βελτίωση της ζωής, για το περιβάλλον, επιτέλους μια κοινωνικονομική αλλαγή και κοινοφελείς υπηρεσίες για να μιλάμε για ένα κοινωνικό πυλώνα. Καν. Πραγματικά με έχει σοκάρει, με έχει συγκλονίσει αυτή η ελαφρότητα, αυτή η επιπολαιότητα, αυτή η αφέλεια και αυτή η ανικανότητα με την οποία χειριζόμαστε τέτοια πράγματα από την πλευρά της Επιτρόπου. Uh, thank you. Ε, Ευχαριστώ. Εδώ τελείωσε ο κατάλογος των ομιλητών μας και θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Πίτροπο για να απαντήσει. Thank you very... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξαιρετικά μέλη, σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις, τις ιδέες, τις ερωτήσεις, τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ενότητες. Ελπίζω να απαντήσω σε όλα τα σημεία. Ίσως να μην ασχοληθώ με το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό, γιατί όπως είπα αυτή είναι μια δοκιμαστική φάση για αυτό το πρόγραμμα, για το επόμενο ε, ΠΔΠ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα το πρόγραμμα των 500 εκατομμύριων, γιατί κάποιος ρώτησε για το πόσα δις. Μιλάμε για 500 εκατομμύρια για μία διετία. 19-20. Θα προσπαθήσω όμως να απαντήσω στις πλήστες ερωτήσεις. Πρώτον, όπως ε, σωστά είπε η κυρία Γκροστέτ, μέχρι στιγμής ήταν θέμα εθνικής κυριαρχίας. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχω παρατηρήσει, ιδιαίτερα στο Συμβούλιο, ε, μια σημαντική αλλαγή. Όλα τα κράτη-μέλη, όλα και τα 28 συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υπέρ, πολύ υπέρ του ε, προγράμματος. Ακόμη και ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, όταν συμμετέχω ε, στη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας, ακόμη και ο Βρετανός εξέφρασε την στήριξή του για το πρόγραμμα αυτό. Όλοι λοιπόν είναι υπέρ του προγράμματος. Αυτό και βέβαια ο μακροχρόνιος στόχος είναι η στρατηγική αυτονομία είναι η ε, γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος, είναι να ανταποκριθούμε σε εξωτερικές και εσωτερικές απειλές. Αλλά στη συζήτηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας ε, των κρατών μελών ανακαλύψαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Όπως είπε και ο κύριος Μποτικόφερ, ε, υπάρχουν προσπάθειες ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά για πρώτη φορά αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που έχουμε πλήρη στήριξη υπέρ της ιδέας και ε, πίσω από αυτό βρίσκεται η δική μας ιδέα για πρώτη φορά να διαθέσουμε ε, κάποια ποσά, όχι πολύ σημαντικά, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να το δοκιμάσουμε. Γιατί ίσως αυτό να κινητροδοτήσει τις επιχειρήσεις. Δεν είναι μεγάλα ποσά για τον τομέα. Δεν είναι κονδύλια που αλλάζουν τα πράγματα και θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις για τον προπολογισμό συγκεκριμένα. Αλλά θα μας δώσει και... Πραγματικά είμαι σίγουρη μετά από τις συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφερόμενους φορείς είμαι σίγουρη ότι αυτό το 20-30% των κονδυλίων θα έχει μεγάλη επίδραση στον τομέα αυτό. Το πιστεύω αυτό. Όπως αναφέρατε, ε, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη, τουλάχιστον δύο εταιρείε που να συμμετέχουν στο έργο αυτό. Το έργο θα πρέπει να συμβαδίζει με τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από τα κράτη-μέλη. Το έργο θα πρέπει να επιλεγεί από την ενισχυμένη πλειοψηφία των κρατών μελών. Γι' αυτό και η συμμετοχή των μικρότερων κρατών μελών ελπίζουμε να εξασφαλιστεί προσπαθώ σε αυτό το σημείο να βλέπω τα πράγματα πραγματιστικά όσο είναι δυνατόν. Βέβαια, έγιναν δύσκολε επιλογέ για τον προπολογισμό, σύμφωνα με τον προπολογισμό. Αλλά μπορώ να σα πω ότι είμαι πολύ ε, σίγουρη ότι αυτέ οι προτινόμενε ε, διαθέσει δεν θα επηρεάσουν την καλή υλοποίηση του προγράμματο. Ο κύριο Μπουτικόφερ αναφέρε ε, κάποια προγράμματα για τα οποία είμαι υπεύθυνη, Γαλιλαίο και Κοπέρνικος. Πιστεύετε ότι θα μπορούσα εγώ να βλάψω τα δικά μου έργα? Όχι. Γι' αυτό υπάρχουν λίγες γραμμές προπολογισμού και λίγα περιθώρια, δεν υπάρχουν πολλά. Ε, δεν ε, πάει πάνω από το 10% του περιθωρίου. Υπάρχουν λοιπόν λιγοστά 1, 2, 3, 4, 5 σημεία όπου προσπαθούμε να συλλέξουμε ε, τα κονδύλια. Συζητάμε, ε, συζήτησα με τους συναδέλφους επιτρόπους και βέβαια οι περιορισμοί του προπολογισμού είναι γνωστοί ε, σε όλους. Αλλά θα πρέπει να βρούμε μια λύση σε αυτό το πλαίσιο και ελπίζω να βρεθεί ένας καλός συμβιβασμός σε αυτό το σημείο, γιατί πιστεύω και είμαι σίγουρη ότι το αξίζει, αξίζει να γίνει αυτό, ε, και για τον οικονομικό αντίκτυπο της αμυντικής βιομηχανίας. Υπάρχουν εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, ε, το μέλλον ε, του ΑΕΠ για κάποια κράτη-μέλη, μεγάλη αξιακή αλυσίδα για πολλά κράτη-μέλη. Αυτές είναι γραμμές πάνω στις οποίες μελετούμε το θέμα και προτείνουμε βέβαια να περιορίσουμε τη χρηματοδότηση μόνο σε ευρωενωσιακές εταιρείες. Γι' αυτό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δύο κριτήρια της τοπικοποίησης, ε, όπως και με την προπαρασκευαστική ε, δράση, να υπάρχουν οι ε, οι εγκαταστάσει υποδομή να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο αποτελεσματικό έλεγχος που θα καθορίσει την κυριότητα, 50%. Αυτό το κριτήριο της κυριότητας, της διοκτησία του 50% έχει επικριθεί. Είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, αλλά γι' αυτό ε, αυτό είναι ο ρόλος σας, να προτείνετε κάτι. Δεν λέω ότι εγώ ε, τα έχω, όλες τις λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Θέλουμε να ε, πετύχουμε την καλύτερη δυνατή επίδραση για να έχουμε την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όλων των κρατών μελών. Δεν είμαι υπέρ του georeturn, return Ίσως να πω ε, δύο λόγια στα πολωνικά. Ναι, γιατί αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη, και μεγάλα και μικρά. Αναφερθήκατε σε μεσαίου εταιρείε. Εμείς μιλάμε για μεσαίου μεγέθους εταιρείε. Αυτές οι εταιρείε στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν στον αμυντικό τομέα, στον τομέα της άμυνας. Δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες εταιρείε, αλλά μεσαίου μεγέθους εταιρείε. Και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε όλες αυτές τις εταιρείε και όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιδείξουν ενδιαφέρον σε αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό ισχύει και για τις εταιρείε. Οι εταιρείε θα πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον. Θα κάνω μια περιοδία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης για να συναντήσω εταιρείε. Θα μεταβώ σε κράτη-μέλη, όχι στα μεγαλύτερα κράτη-μέλη, αλλά σε εκείνα τα οποία έχουν έναν τομέα άμυνας για να μοιραστώ μαζί τους και να μεταδώσω όλες αυτές τις πληροφορίες και να βεβαιωθώ ότι οι εταιρείε έχουν πρόσβαση στις βέλτιστες καλύτερες πληροφορίες και για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείε και για αυτές που δεν συμμετείχαν ήδη σε ένα τέτοιο έργο είναι ε, θετικό. για τις εταιρείες που δεν είναι ευρωπαϊκές και τις βρετανικές εταιρείε. Υπήρχαν δύο ερωτήσει γι' αυτό. Τις μη Ευρωπαϊκέ και βρετανικέ εταιρείε, Όπως είπα, τα ωφέλη του προγράμματος είναι ε, για επιχειρήσεις που βρίσκονται, που είναι εγκαταστημένες στην Ένωση. Οι επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια τώρα μπορούν να υποφελούνται. Αλλά οτιδήποτε άλλο εξαρτάται από τι διαπραγματεύσει και μεταξύ του Μισελ Μπανιέλ και του Ντέβιτ Σιλ. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Άκουσα όμως επανειλημμένος ε, τον Υπουργό, τον Βρετανό, να είναι υπέρμαχο του προγράμματος αυτού ε, για 60 χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εναντίον σε οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Τώρα είναι πολύ υπέρ του προγράμματος αυτού. Τώρα, για τον ορίζοντα 2020 στην ε, ανακοίνωση που συνοδεύει το πρόγραμμα το καταστήμα σαφές ότι το μελλοντικό ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να είναι διαχωρισμένο σαφώς από το FP9. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, τους κανόνες, τις διαδικασίες. Ελπίζω αυτό να ανταποκρίνεται στη συζήτηση και να είναι σαφές. Τώρα για, την, το ΠΕΣΚΟ, τη μόνιμη διαθρωμένη συνεργασία, ήταν ερώτηση του κ. Κρασναντένσκι. Το πρόγραμμά μας είναι ξεχωριστό από την ΠΕΣΚΟ. Όμως έγιναν εκκλήσεις και αιτήματα από κράτη-μέλη να κάνουμε μια διασύνδεση, ένα σύνδεσμο με αυτό. Δεν θέλαμε να το κάνουμε, αλλά σε κάποια περιορισμένα έργα γιατί βέβαια δεν είναι όλα τα προγράμματα ΠΕΣΚΟ που θα ε, εμπίπτουν. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε να κάνουμε μόνο για τεχνολογικής φύσεως προγράμματα και έργα. Αλλά εκεί θα διαβουλευτούμε με τα κράτη-μέλη και αποφασίσαμε να αυξήσουμε τη συγχρηματοδότηση στο 30%. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη τι είδους προγράμματα ΠΕΣΚΟ θα προταθούν. Δεν παρεμβαίνω με κανένα τρόπο σε αυτή τη διαδικασία, αλλά το ΠΕΣΚΟ θεσπίστηκε και πολλές φορές αυτό έχει θίξει ε, και ο Πολωνός Υπουργός Άμυνας ότι θα πρέπει να, κάποια, να υπάρξει κάποια σύνδεση. Για την νομική βάση ήθελα να το αφήσω στο τέλος αυτό το σημείο της νομικής βάσης. Θα πω ότι κατανοώ τις απόψεις σας και συμμερίζομαι την απόψη σας, αλλά εμείς ε, το αναλύσαμε από νομικής άποψης, εις βάθος το θέμα. Εξετάσαμε προσεκτικά διαφορετικές νομικές λύσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η νομική βάση το 173 είναι μια γερή νομική βάση που να ανταποκρίνεται στους στόχους του προγράμματος. Αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται κάποια πολιτική βάση. Αυτά τα δύο άρθρα, το 254 και 255, όπως τα έχουμε εμείς εξετάσει δεν αποτελούν αυτά καθ' αυτά μια νομική βάση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νομική βάση ακόμη και αν σχετίζονται με το άρθρο 173. Για την ώρα λοιπόν, μετά από ενδελεχή νομική ανάλυση αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το άρθρο. Εάν υπάρξει η πιθανότητα δεν ακούγονται τα σχόλια, σχόλια εκτός μικροφώνου. Επίτροπος. Δεν μπορώ να δεσμευτώ, αλλά θα το ελέγξω, θα το, θα το δω. Θα το κοιτάξω το θέμα. Έχουμε μιλήσει για τις μικρομεσές. Νομική ανάλυση το καλύψαμε. Τώρα, τα τελευταία δύο σημεία. Πρέπει να δημιουργηθεί μια συνεργασία στον τομέα. Μέχρι στιγμής γίναν κάποιες δοκιμές, αλλά τώρα έχουμε αυτό το momentum και είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει. Προσπαθούμε λοιπόν με περιορισμένα κονδύλια και βεβαίως όπως σας είπα και προηγουμένως πριν από τρία χρόνια όταν το ξεκινήσαμε όταν ανέλαβα δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι σε 18 μήνες θα μπορούσαμε να κάνουμε τόση πρόοδο στην συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Θα προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ρεαλιστές μπορούμε με περιορισμένα κονδύλια, ξεκινώντας με την έρευνα, προχωρώντας στη συνέχεια με τις ε, δυνατότητες, το μέρος που έχει να κάνει με τις ικανότητες και αυτό προτείνουμε. Βέβαια, είμαι ανοιχτή σε εισηγήσεις, προτάσεις, παρατηρήσεις, αλλά νομίζω βλέπετε το πώς το βλέπουμε κι εμείς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει το 2019. Εάν όχι, τότε η πρόταση δεν θα ισχύει πια. Δεν θα έχει ενδιαφέρον για τα κάτι μελη Και ήθελα να τονίσω επίσης ότι η Εστονική Προεδρία έχει δεσμευτεί σχεδόν ότι θα έχει μια γενική προσέγγιση μέχρι τον Νοέμβριο, τον επόμενο μήνα. Θα πρέπει να επιταχύνουμε λοιπόν τη διαδικασία και θέλω να στηρίζομαι σε εσά και στη στήριξή σας. Τώρα, σχετικά με την βιομηχανική στρατηγική. Ο κύριε Μαρτά, σίγουρα ξέρετε ότι συμμερίζομαι τις απόψεις σας για τους κανόνες του ανταγωνισμού. Και ε, οι κανόνες του ανταγωνισμού θα πρέπει να έχουν σφαιρική παγκόσμια ε, διάσταση, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα σφαίροντα των ενδιαφερομένων ε, μερών και τα συζητάμε εδώ και κάποιους μήνες στην Επιτροπή. Προσπαθώ να αλλάξω την προσέγγιση στην ίδια την Επιτροπή. Γιατί συμφωνώ για αυτό το θέμα του ανταγωνισμού, για τον φόρο ε, για τον άνθρακα. Είναι μια δυνατότητα να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην παρέμβουμε με τους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους μας όπως είναι είπα και η Κίνα, αλλά συνεχίζονται οι συζητήσεις στην Κομισιόν με αργούς ρυθμούς μεν, αλλά ε, ακόμη συζητούνται και μέχρι στιγμής έχουμε ε, δώσει ε, είμαι έτοιμη να το ε, εξετάσω και αυτό μπορώ να σας πω επίσης ότι έχουμε συνεχιζόμενη πρωτοβουλία στον κύριο και έχουμε μια συνεχιζόμενη πρωτοβουλία για τα μέταλλα και τις πρώτες για να μειώσουμε την εξάρτηση από εισαγωγές από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες. Συζητάμε επίσης το θέμα αυτό στην θέμα της κυκλικής οικονομίας και αυτό είναι επιτάπητος και συζητείται στην Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Επίτροπε. Πολύ ενδελεχή συζήτηση. Όλες οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη με κάποιο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι 100% πάντα, γιατί είναι και αδύνατον, αλλά κάποιες από αυτές μπορεί να επηρεάσουν την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως υπάρχει ε, μια γενική υποστήριξη και στους ευρωβουλευτές ε, προς το πρόγραμμα, όχι μόνο από τα κράτη-μέλη, έτσι. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, όλες οι προτάσεις σας, όλες οι αφιβολίες σας, όλα σας τα σχόλια είναι σημαντικά. Τελειώνουμε και εγκαίρος μάλιστα σήμερα. Έχουμε τρία λεφτά ακόμα. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Δεν νομίζω. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα. Θα τα ξαναπούμε στις 11 και 12 του μηνός. 11 και 12 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα.